Right, good morning. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινούμε σήμερα τη συνεδρίαση με την παρουσίαση των τριών μελετών για την εφαρμογή τη Συμφωνίας σύνδεση με τη Μολδαβία, τη Γεωργία και την Ουκρανία. Πριν να περάσουμε στην πρώτη παρουσίαση από των, εκθέσεων που έχουν καταρτιστεί από τους κυρίους Τρεβίτσιους, Μαμίκινς και Γκάλερ. Αυτές οι μελέτες ε, παρέχουν ε, εις βάθος εμπειρογνωμοσύνη στην Επιτροπή μας ε, εν ώψη της εργασίας μας για τις τρεις εκθέσεις και συμπληρώνουν την εμπειρογνωμοσύνη που αποκτήσαμε πέρσι με τη μελέτη για την εκλογική μεταρρύθμιση στην ε, περιοχή, τι συνεισφορέ τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τη Κομισιόν και τι ερευνητικέ αποστολέ τη Επιτροπή μα. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε οι εμπειρογνώμονε να μα δώσουν κάποια περαιτέρω στοιχεία για την πρόοδο που έχει γίνει ε, για τις σχέσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση των εταιρών αυτών και να μας προτείνουν κάποιες ξεκάθαρες συστάσεις πολιτικής. Γι' αυτό τους έχουμε καλέσει για να μας παρουσιάσουν τις μελέτες τους ε, Καμίλ Κάλους που θα παρουσιάσει την ε, εφαρμογή της συμφωνίας με τη Μολδαβία. Καλωσορίζουμε στη συνέχεια την Όνα Μικελίτσα από τη Γεωργία θα μας παρουσιάσει τη δεύτερη μελέτη που αφορά την εφαρμογή τη Συμφωνία Σύνδεση με τη Γεωργία και τον ε, δόκτωρ Άντρε Τούσκα που θα μας παρουσιάσει την εφαρμογή της συμφωνίας με την Ουκρανία. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονες και να τους δώσω το λόγο για 10 λεπτά ο καθένας. Ε, μπορείτε να μιλήσετε και στη συνέχεια θα περάσουμε στη συζήτηση. Ξεκινάμε με εσά, κύριε Κάλλους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε και κύριοι. Θα περιοριστώ στα κυρία απορίσματα και ευχαρίστω ε, να απαντήσω στις ερωτήσεις. Ε, αυτές ε, οι μελέτες είναι μέρος ε, της Ευρωπαϊκής Μελέτης Αξιολόγησης. Ας ξεκινήσουμε με τα απορίσματα και τα συμπεράσματα. Το συνολικό αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν στη Μολδαβία μεταξύ του 2014 και 2018 θα πρέπει να αξιολογηθεί ως μη ακονοποιητικό. Έχαμε σταδιακή επιδείνωση των δημοκρατικών μηχανισμών, κυρίως τα δύο τελευταία με τρία χρόνια. Επίσης, η Μολδαβία ε, θεωρεί το 2016-2017 ως ένα κράτος όπου κυριαρχούσε ο κύριος Πλατχόνιουκ, ο οποίος ε, είναι ολιγάρχης και επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος. Ε, βέβαια, η πρόοδος που σημειώθηκε δεν συνοδεύτηκε από πολιτική πρόοδο. Έχουμε μία βελτίωση τη νομική και θεσμική βάση στην Μολδαβία, αλλά η κατάσταση σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου, την καλή διακυβέρνηση και τη δικαιοσύνη ιδίω και των δημοκρατών κρατήτων, είτε δεν σημείωσαν σημαντική βελτίωση ή σημειώνονται πιστοδρόμηση. Τα προβλήματα επίση είναι ότι οι κανονισμοί δεν εφαρμόζονται παρκώ, κάποιε μεταρρυθμίσει ε, ε, έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των κυβερνώντων, επομένω ε, δεν υλοποιούνται. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κύρια απορίσματα, θα ξεκινήσουμε με το σύστημα της δικαιοσύνης που παραμένει ε, ένα, ένας από τους τομείς όπου έχει υποστεί τις λιγότερες μεταρρυθμίσεις. Ε, παραμένει το δικαστικό σύστημα ιδιαίτερα διεφθαρμένο και δείχνει μία ε, στάση υπηρετική προς τις πολιτικές επιχειρηματικές ομάδες. Επίσης, συχνά χρησιμοποιείται από τον πλατχόνιο και το δικαστικό σύστημα κατά των ε, πολιτικών του αντιπάλων και ε, είδαμε ότι τους ε, τελευταίους μήνες είχαμε και επίθεση κατά των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, επίσης, ένας από τους ε, κυρίους ε, λόγους για την έλλειψη πρόοδου στην έρευνα για την κλοπή του ενός δισεκατομμυρίου είναι η πολιτική εξάρτηση του δικαστικού σώματος. Η κυβέρνηση έχει αναγκάσει το δικαστικό σώμα να υπακούει σε αυτή, χρησιμοποιώντας διάφορες τακτικές εκφοβισμού. Τώρα, το συνταγματικό δικαστήριο παραμένει ιδιαίτερα πολιτικοποιημένο. Οι αποφάσεις ε, είναι, ε, έχουν πολιτικά κίνητρα και ουσιαστικά μερικοί έχουν αλλάξει κάποια κύρια στοιχεία του πολιτικού συστήματος της Μολδαβίας, ε, μην ακολουθώντας την κλασική νομοθετική οδό η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει κάνει καμία ουσιαστική προσπάθεια να αυξήσει την ανεξαρτησία ε, του συνταγματικού δικαστηρίου. Τώρα, τα θετικά στοιχεία υπάρχουν ε, κάποια απορίσματα που είναι κάπως αισιόδεξα. Τον Νοέμβριο του 2017 πρότεινε η κυβέρνηση μια σειρά μεταρρυθμίσεων στο Σύνταγμα που θα πρέπει να αυξήσει την ανεξαρτησία των δικαστών. Ωστόσο, ο νέος κανονισμός δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα. Επίσης, ο κωδικός αστικής ε, δικονομίας τροπήθηκε τον Απρίλιο του 2018 προκειμένου να μειωθεί ε, η διάρκεια των δικών, απλουστεύοντας τις διαδικασίες και το Μάρτιο του 2017 θετήθηκε εθνική ε, στρατηγική κατά της διαφθοράς. Σε ό,τι αφορά τώρα την καταπολέμηση της διαφοράς, ε, όπως σας είπα στην αρχή, η νομική βάση έχει βελτιωθεί, αλλά η πολιτική εξάρτηση και περιορισμένη αποτελεσματικότητα αυτού του θεσμού παραμένει προβληματική. Θεσμοί όπως το Εθνικό Κέντρο Καταπολέμησης της Διαφθοράς παραμένει πολιτικοποιημένο και δεν είναι αποτελεσματικό, ε, καθώς προβαίνει σε καταχρήσεις, ε, η ανεξαρτησία ε, του εισαγγελέα και της διαφθοράς ε, αμφισβητείται. Ε, σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες παραμένει ο θεσμός αυτός υπό τον άμεσο έλεγχο του Βλάτ Πελατχόνιουκ. Ένα άλλο αρνητικό είναι ότι η Εθνική Αρχή Ακαιρεότητας που δημιουργήθηκε το 2016 δεν έχει λειτουργήσει μέχρι το Φεβρουάριο του 2018 όταν το Κοινοβούλιο τελικά ενέκρινε την δομή της, ε, την οργανωτική δομή του θεσμού. Επίσης, ε, κάτι θετικό, έχουμε την υιοθέτηση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της, ε, του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος και της τρομοκρατίας και το πλαίσιο των μέτρων κατά της διαφθοράς που επικαιροποιήθηκε το Μάρτιο του 2017. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει επαρκή πρόοδος στην καταπολέμηση της διαφθοράς ε, και αυτό έχει εκδοτηθεί στη μασκοπήση. Το 96% των Μολδαβών πιστεύουν ότι είναι πολύ μεγάλο θέμα η διαφθορά και φυσικά δεν μειώνεται, δυστυχώς δεν μειώνεται αυτός ο αριθμό, αλλά αυξάνεται συνεχώς. Λοιπόν, για την απάτη του ενός δισεκατομμυρίου. Η έρευνα αυτής της υπόθεσης ε, δεν έγινε αποτελεσματικά. Μέχρι σήμερα οι αρχές δεν, ε, δεν έχουν μπορέσει να ανακτήσουν ε, κανένα ποσό και έχουν επιστρέψει περίπου 50 εκατομμύρια, αλλά αυτά δεν είναι από τα κλαμμένα χρήματα. Αυτά είναι χρήματα που προέρχονται από την πώληση των χρημάτων ε, σε μια τράπεζα. Η πλήρης ε, εκδοχή τη δεύτερη εκθέση Κρόλ δεν έχει δημοσιευτεί και τον Ιούνιο του 2017 ο Ιλιαν Σόρ, ο πολιτικό και επιχειρηματία που θεωρείται ότι είναι ο κύριο αρχιτέκτονα τη απάτη, καταδικάστηκε σε 7,5 χρόνια κάθυρξη, αλλά σήμερα ε, είναι υποδικαστικό έλεγχο και περιμένει την τελεσίδικη απόφαση του εφετείου και είναι πάρα πολύ ενεργός πολιτικά και επιχειρηματικά και μπορεί και εύκολα να φύγει από τη χώρα το επιθυμεί. Τώρα, να σας ε, πω ποια είναι τα απορίσματα και τα συμπεράσματα. Καταρχήν, τους τελευταίους πολλούς μήνες έγινε προσπάθειες να περιοριστεί η ελευθερία της δράσης ε, των ε, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και να απαξιωθούν ε, στα μάτια του κοινού. Ιδιαίτερα το είδαμε αυτό τον τελευταίο καιρό, μεταξύ του 2016 και 2018, η σύλληψη και περικοπή των πολιτικών αντιπάλων ήταν πολύ πιο συχνή, παρά την εισαγωγή ενό νέου νόμου για την μονοπόλιο των ΜΜΕ, αυξάνεται το μονοπόλιο στα χέρια των ε, κυβερνώντων ε, και επίσης έχουμε όλο ένα και περισσότερο εκφοβισμό των δημοσιογράφων. Η πολιτική πίεση στις τοπικές αρχές και ο εκφοβισμός των εκπροσώπων τους από τις αρχές είναι κάτι κοινό. Σύμφωνα με τα δεδομένα, περίπου 20%, 21% των εκπροσώπων των τοπικών αρχών έχουν ε, δεχτεί απειλές σωματικές ή ψυχολογικές και το 15% έχει χάσει τη δουλειά του και αυτά είναι δεδομένα του 2018. Η νομική βάση, και αυτό είναι κάτι θετικό, στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει βελτιωθεί κατά την περίοδο πανελίου, αν και κάποιες ελλείψεις ε, στη διαδικασία της υιοθέτηση παρατηρήθηκαν. Δυστυχώ, άδικε δίκε εξακολουθούν να υπάρχουν στη Μολδαβία. Κάποιε μηνύσει ε, χωρί αποδεκτικά στοιχεία κατατίθενται κατά των πολιτικών, την των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Οι αλλαγές του εκλογικού συστήματος ε, που υλοποιήθηκαν το δεύτερο ήμιση του 2017 ε, ουσιαστικά ευνόησαν το κυβερνών ε, κόμμα αλλά και το σοσιαλιστικό κόμμα και παραβίασαν τις διεθνείς συστάσεις και πρότυπα αλλά και τους εγχώριους νόμους. Ε, περιπτώσεις σοβαρών περιορισμών του δημοσίου δικαιωμάτως να συμμετέχει στην διαδικασία λήψης αποφάσεως παρατηρήθηκαν πρόσφατα Επίσης είδαμε τι συνέβη και με τα εκλογικά αποτελέσματα ε, στην εκλογή του Δημάρχου του Κισινάου θετικό. Η εφαρμογή της DCFTA όθεσε το εμπόριο Μολδαβίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 2015-2017. Αυξήθηκαν και εξαγωγές και εισαγωγές κατά 31 και 22% αντίστοιχα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε ο κύριος εταίρος της ε, χώρας, ε, ο κύριος εμπορικός εταίρος ε, και ο μεγαλύτερος επενδυτής για την περίοδο 2014-2016. Το 2017, 66% των συνολικών εξαγωγών πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με το 47% το 2013. Οι μεταρρυθμίσει ε, στον ε, χρηματοπιστωτικό τομέα συνεχίζονται και θεωρήθηκαν ότι είναι θετικές. Ε, όμως η έρευνα για την τραπεζική απάτη είναι το κύριο πρόβλημα, η κυρία παράληψη της κυβέρνησης και δυστυχώς βλέπουμε έναν αργό ρυθμό θεσμικών μεταρρυθμίσεων και αυτό θέτει σε κίνδυνο τις θετικές αλλαγές στην οικονομία. Θα σταματήσω εδώ νομίζω γιατί μου τέλειωσε ο χρόνος και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε. Ακριβώς στα 10 λεπτά, αλλά βέβαια μιλήσατε πάρα πάρα πολύ γρήγορα, έτσι. Συγγνώμη, David. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει να, να ακούσουμε και τις τρεις παρουσιάσεις και μετά οι ερωτήσεις και τα σχόλια. Ε, να στρέφονται, δεν ξέρουμε κι εμείς σε ποια από τις τρεις. Οπότε καλύτερα είναι να γίνει πρώτα ένας γύρος ερωταπαντήσεων και μετά να περάσουμε στις επόμενες. Γιατί μετά κάπως θα τα μπλέξουμε. Εντάξει, ο Μιχαλ Γκάλερ αυτό πρότεινε, τι λέτε κι εσείς, συμφωνείτε. Ωραία, συνολικά για αυτές τις τρεις μελέτες έχουμε μία ώρα. Ωραία. Έχουμε λοιπόν 10 λεπτά για τη Μολδαβία. Ερωτήσεις. Παρακαλώ. Θα έρθει και σας η ώρα σας μετά. Η Σάντρα πρώτα. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω λετωνικά. Παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας. It's fine. Nesen notikušo vietējo vēlēšanu ε, ακυρώθηκε το αποτέλεσμα στις τοπικές εκλογές και υπάρχει μια συνεχής ε, πίεση στον ηγέτη της αντιπολίτευσης. Γεγονός που μας ανησυχεί η ακύρωση του αποτελέσματος δείχνει ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη και ότι οι ολιγάρχες έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Η απάτη του ενός δισεκατομμυρίου δεν έχει ενόχους. Έγινε μια δίκη υπέφερε η κοινωνία των πολιτών από αυτή. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η οικονομική ενίσχυση, η μακροοικονομική ενίσχυση μετά τις ε, κοινοβουλευτικές εκλογές και μόνο υπό την προπόθεση ότι οι εκλογές θα πληρούν τα διεθνή πρότυπα. Α, πολύ χαρήκαμε που σας ακούσαμε να μιλάτε λετωνικά. Πέτερς. Ευχαριστώ, David. Να ξεκινήσω λέγοντα ότι ήταν ε, μια πολύ ορθή απόφαση της Επιτροπής μας ε, να παραγγείλει αυτές τις εκθέσεις από αυτούς τους ε, εξαιρετικούς εμπειρογνώμονες που έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα. Άκουσα, ε, συγγνώμη, διάβασα το κομμάτι που αφορούσε τη Μολδαβία σαν να ήταν μυθιστόρημα. Ήταν πολύ περιεκτικό, ακριβές και πραγματικά σας συγχαίρω για το έργο σας. Η σύνοψη που μας παρουσιάσετε είναι εξαιρετικά σαφής. Δυστυχώς δεν είναι πολύ θετική ως προς ε, ε, την άρχουσα τάξη της ε, την, την ελίτ που διοικεί τα πραγματική. Αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να ρωτήσω τα εξής. σε ό,τι αφορά τα ευρήματά σας. Τι περιμένετε από την εισαγωγή αυτού του μικτού εκλογικού συστήματος. Οι εκλογές αναβάλλονται για τα τέλη Φεβρουαρίου του 19. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το αποτέλεσμα μετά από αυτό τον κοινωνικό στοχασμό ή προβληματισμό, αν θέλετε. Και δεύτερον, στα τέλη Ιουλίου το Κοινοβούλιο της Μολδαβίας υιοθέτησε ένα πακέτο για τη φορολογία που ουσιαστικά ε, δίνει ελαφρύνσεις ε, κεφαλαϊκές. Τι αναμένεται από αυτό. Οι πρώτες ε, αντιδράσεις από τη Δύση ήταν πολύ αρνητικές. Ευχαριστώ. Claire Moody. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την έκθεση και για όλη τη δουλειά που κάνατε. Ένα πολύ απλό ερώτημα από πλευρά μου. Ποιες είναι οι συστάσεις σας προς εμάς μετά τα όσα έχετε δει σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας ε, με τη Μολδαβία και στο πλαίσιο βέβαια της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης. Ευχαριστώ, Μιχαήλ, τέλος. Θα μιλήσω και εγώ γερμανικά. Υποστηρίζω την επιθυμία της Άνδρα Καγέτο να έχουμε μια αυστηρή αιρεσιμότητα ως προς ε, την ε, μακροοικονομική οικονομική ενίσχυση με έχει εξοργήσει η εξέλιξη εκεί και θα πρέπει να εστιάσουμε σε δύο τομείς ενάντια στις συμβουλές και σύμφωνα με την Επιτροπή της ε, Βενετίας υπάρχει ένα ανορθόδοξο εκλογικό σύστημα όπου υπάρχει μισή εξουσία από δύο διαφορετικά κοινοβούλια ουσιαστικά ώστε να έχει επιρροή ο ολιγάρχης. Θεωρώ ότι αυτό το σύστημα δεν είναι κατάλληλο. Δεν θα κερδίσουμε τίποτα από ένα τέτοιο σύστημα, ένα τέτοιο αναλογικό. Θεωρώ ότι δεν θα εξυπηρετήσει σε τίποτα κάτι τέτοιο. Προσπαθήσαμε λοιπόν στην ε, αρχή του τελευταίου χρόνου μαζί με δύο ιδρύματα, ο Κόναντα να Αστίφτουν και ένα ακόμα, να προειδοποιήσω ότι αυτό το εκλογικό σύστημα είναι λάθος να το εφαρμόσουμε. Παρ' όλα αυτά έγινε. Κατά την άποψή μου. Ακόμα χειρότερη είναι η συμπεριφορά μετά τις ε, δημοτικές εκλογές στην πρωτεύουσα, όπου κέρδισε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης θεωρώ ότι είναι σύμφωνα όλα αυτά που συνέβησαν ε, με την μελέτη ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη. Είναι καταστάσεις που δεν πρέπει να δεχόμαστε. Και επομένω, αν δεν αλλάξει η κατάσταση, δεν είμαι πρόθυμος να συνεχίσω και να υποστηρίξω τη συνέχιση των, της οικονομικής ενίσχυσης. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Έχουμε... Ο κύριος Ζωσνιέτς, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ. Και πάλι βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υιοθετεί ψήφισμα για τη Μολδαβία και μπαίνει σε δύσκολη θέση. Ουσιαστικά μιλάμε για την αγυρότητα των εκλογών, αλλά και τι θέλουμε τελικά. Ε, στην Πολωνία ε, την επικρίνουμε επειδή αλλάζει το σύστημα, τη Μολδαβία την επικρίνουμε επειδή δεν το αλλάζει. Τι συμβαίνει τελικά και τι θέλουμε. Any request to speak not... Δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Όχι. Πέντε ομιλητές, αρκετές ερωτήσεις. Σε πέντε λεπτά να απαντήσετε παρακαλώ. Ναι, θα τα καταφέρω, πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και τα σχόλια. Το πρώτο είναι και το πιο σημαντικό. Τι μπορούμε να περιμένουμε μετά τις εκλογές του Φεβρουαρίου. Και εμείς αυτό διερωτώμεθα και δεν έχουμε κάποια καλή απάντηση να σας δώσουμε. Η απόφαση αναβολής ε, των εκλογών για το Φεβρουάριο προέκυψε από το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών στο Κισινάου, το οποίο και οι αρχές οι ίδιες το εξέτασαν ως μια δοκιμασία. Ήθελαν να δουν αν θα λειτουργήσει το σύστημα και αν θα κατάφεραν να περάσουν τους υποψηφίους. Τελικά όχι. Οπότε χρειάζονταν περισσότερο χρόνο. Γι' αυτό και πήγαμε το Φεβρουάριο. Από την άλλη έπρεπε κάπως να καλύψουν αυτή την κακή εικόνα των αρχών μετά από αυτή την ε, απόφαση. Γι' αυτό η οποία απόφαση έτυχε δρυμύτα της κριτικής, για να απαντήσω και στο τελευταίο ερώτημα. Νομίζω ότι η αλλαγή του δικαστικού συστήματος και η μεταρρύθμιση του θα βοηθούσε ε, να λάβουν μεγαλύτερη στήριξη οι δημοκράτες από ό,τι συνήθως. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά το πάγωμα της μακροοικονομικής βοήθειας. Υπήρξε λοιπόν επιστολή από πάνω από 700 ε, δημάρχους ε, στη Μολδαβία, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική εξάρτηση ε, των τοπικών αρχών από τις κεντρικές και αυτό σίγουρα αξιοποιείται και στις εκλογές. Σίγουρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Από την άλλη πιστεύω ότι θα υπάρξει ένας ε, τυπικός ή άτυπος ε, συνασπισμός μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν βλέπω άλλη επιλογή. Ίσως θα μπορούσε να υπάρξει συνασπισμός μεταξύ της φιλοευρωπαϊκής ε, αντιπολίτευσης και των δημοκρατικών, αλλά βέβαια με τη στήριξη του κυρίου Μπαχατιούκ, όμως αυτό δεν γίνεται πια με, με τη σχέση των, ε, των όσων ελέγχουν τα μέσα σε σχέση με την αντιπολίτευση. Κατά λοιπά δεν έχω πολλά να προσθέσω ε, στα όσα έχουν πει οι διεθνείς οργανισμοί και η ΜΚΟ στη Μολδαβία που έχουν επικρίνει δρυμύτατα τον νέο νόμο. Κατανοητό το σκεπτικό βέβαια, του νόμου και τελικά και ο κύριος Ντοντών τη στήριξε. Στήριξε τον νόμο. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα πολιτικό καρτέλ στη Μολδαβία. Συστάσεις τώρα. Κάποια σίγουρα συμπεριλαμβάνονται και στην έκθεση. Όμως το πιο σημαντικό, παρότι ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, είναι να είμαστε ακόμα πιο αυστηροί και σκληροί ως προς την κυβέρνηση. Αν δείτε και τις δημοσκοπήσεις μετά το πάγωμα της μακροοικονομικής ε, ε, στήριξης, θα δείτε ότι η στήριξη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να αυξάνεται. Μπορεί να ήταν μόνο λίγες ποσοστιαίες μονάδες, αλλά κάτι άλλαξε, γιατί είδαμε ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε κάτι να κάνει. Ε, οι περισσότεροι δεν πίστεψαν το αφήγημα της κυβέρνηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει τα χρήματά μας από τα σχολεία και τα μα. μας. Ε, κάτι το οποίο είχε πει ο Πρωθυπουργό τη Μολδαβίας. Αυτό είναι το ένα. Μετά, καλό θα ήταν να επικεντρωθείτε περισσότερο προς ε, μεταρρυθμίσεις με γνώμονα τον άνθρωπο και όχι τους θεσμούς γιατί υπάρχει η γενικότερη αίσθηση στη Μολδαβία ότι η οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάει κατευθείαν στις τσέπες ε, της άρχουσας τάξης. Και για το τελευταίο ερώτημα, εν μέρη το απάντησα, συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει παράνομα πράγματα. Στην περίπτωση της Μολδαβίας, δεν γίνεται να αντιμετωπίζουμε την δικαστική απόφαση για την ακύρωση των εκλογών χωρίς ε, να εξετάζουμε το ευρύτερο πλαίσιο, την ευρύτερη κατάσταση στη χώρα. Χωρίς να βλέπουμε πώς αυτή η χώρα άλλαξε τα τελευταία χρόνια, πώς οι θεσμοί ε, ελέγχονται πλήρως από συγκεκριμένα άτομα. Και αυτό το έχω αναφέρει και στην έκθεση και στην ε, ανάλυση που κάνω καθημερινά. Τα πράγματα δεν είναι ίδια με την Πολωνία, κατά οποιονδήποτε τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κάλους, σας ευχαριστούμε για την ε, ανάλυση που κάνατε της κατάστασης στη Μολδαβία. Πολλοί από τους συναδέλφους ε, συμμερίζουν την απόψή σας ότι η χώρα ε, διάγει μία και διανύει μια μεγάλη πολιτική κρίση, το οποίο συνδέεται και με την αιρεσιμότητα στη μακροοικονομική βοήθεια. Για πρώτη φορά, νομίζω, τουλάχιστον σε αυτή την ε, θητεία, εξετάζουμε το θέμα της Μολδαβίας χωρίς καμία συμμετοχή Ρουμάνων συναδέλφων. Συνήθως όταν ε, τίθεται το θέμα της Μολδαβίας ε, στη μέσα διάταξη εμφανίζονται και οι Ρουμάνοι, αλλά όχι σήμερα. Αυτό είναι μια νέα εμπειρία για μας. Μπορούμε να περάσουμε τώρα σε μια νέα γεωπολιτική αλλαγή. Να περάσουμε στη Γεωργία. Κυρία Μικελίτσα, για 10 λεπτά. Thank you. Thank you. Ευχαριστώ. Και στην η υπηρεσία ερευνών που μας βοήθησε σε αυτή την έκθεση. Το 2016 η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης από τότε αντιμετωπίζει προκλήσεις η Γεωργία για να μπορέσει να εφαρμόσει αυτή την σφαιρική σε βάθος ζώνη ελευθερών συναλλαγών. Προσπαθούμε να αναλύσουμε διάφορα επίπεδα της εφαρμογή, ε, ειδικά ως προς το πολιτικό κομμάτι και εστιάσαμε στο κράτος δικαίου, την, ε, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, την ελευθερία του τύπου και άλλες μεταρρυθμίσεις στον οικονομικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Το συμπέρασμα είναι ότι η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλες ε, προκλήσεις ως προς το πολιτικό κομμάτι της Συμφωνίας Σύνδεσης. Έχει κάποιες επιτυχίες στην εφαρμογή της DCFTA. Αξιολογήσαμε τις διαδικασίες που μεταρρύθμισης του 2016 για να αναφέρουμε κάποια βασικά συμπεράσματα και λήψεις που αντιμετωπίζουμε με την εφαρμογή, με το πολιτικό κομμάτι της συμφωνία σύνδεση. Πρώτον, η άτυπη κυβέρνηση παρασκηνιακή πολιτική είναι μια μεγάλη πρόκληση για τη δημοκρατία και δείχνει πόσο προπαγής ε, είναι η πολιτική στη χώρα, η βάση του κράτους που έχουμε. Έχουμε σε αυτό παράγοντες ε, μη κρατικού, ρυθμιστικές αρχές και φυσικά κύριε ο αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος ο Ιβάνης Το να συμπεριλάβουμε την κοινωνία καθιστά την κυβέρνηση λιγότερο απειλητική από ό,τι ήταν αυτή του κυρίου Σακιασβίλη, γιατί τώρα έχουν διαφορετικές μεθόδους η δημοκρατική μετάβαση και η επιτυχής μεταφορά εξουσίας του 2012 θεωρείται επιτυχία της γεωργιανής δημοκρατίας, ωστόσο τα χρόνια διακυβέρνηση του κυβερνώντο κόμματο δείχνει ότι οι δημοκρατικές εκλογές δεν σημαίνουν πάντα μια ομαλή μετάβαση προς την δημοκρατία. Αυτή η θεσμή είναι ακόμα αδύναμη και εδώ ερχόμαστε στην επόμενη πρόκληση που είναι ε, το δύσκολο σύστημα ε, ελέγχου του ισολογισμού. Ήταν ένα ε, κράτος το οποίο πάντα κυριαρχούσε ένα κόμμα. Το κυβερνόν κόμμα έχει πλειοψηφία συνταγματική. Η εκτελεστική εξουσία κυριαρχεί πάνω στην ε, κοινοβουλευτική και την ε, δικαστική. Και αυτό σημαίνει ότι η δικαιοσύνη δεν είναι εξάρτητη τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ακόμα πιο αδύναμα, έτσι οθούν τον κόσμο να ψηφίσει το κυβερνόν κόμμα, το Georgian Dream, ή να μην συμμετέχει στις εκλογές. Η ισχύ του Προέδρου είναι περιορισμένη σύμφωνα με το Σύνταγμα. Όλες οι προσπάθειες να ασκήσει ε, βέτο πάντα ήταν αποτυχής. Και τώρα ερχόμαστε στην αχίλιο πτέρνα του πολιτικού συστήματος ε, της ε, Γεωργίας που είναι το δικαστικό. Οι πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί είναι για να διασφαλίσουν την αναξαρτησία, την αμεροληψία, την επαγγελματισμό των δικαστών και το δίκαιο σε μια δίκαιη δίκη. Πιο σοβαρά προβλήματα υπάρχουν σε δύο, βασικές, σε δύο βασικούς είναι η ανεξάρτητη και αποτελεσματική έρευνα, καθώς και το καθεστώς και δικαιώματα των θυμάτων ε, στις ε, ποινικέ δίκες, η δικαστική εξουσία ε, είναι υπό πολιτική επιρροή ομάδων ενδιαφερόντων. Το γραφείο του Συγγελέα θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητο από κάθε πολιτική επιρροή αλλά ε, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θεωρούν ε, ότι η εισαγγελία δεν είναι ανεξάρτητη και επιπλέον οι διαδικασίες επιλογής και διορισμού και εξελόγηση των δικαστών είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Another μια άλλη δυσκολία έχει να κάνει με την αποκεντροποίηση. Αποκέντρωση. Είναι δύσκολο να εφαρμοστούν οι στόχοι για την αποκέντρωση. Αντίθετα, το 2017 το Κοινοβούλιο ε, έκρινε ένα νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας και μείωσε το θέμα των, αριθμών των αυτοδικούμενων πόλεων από 12 σε 5 με τη δικαιολογία ότι θέλει να αυξήσει την αποδοτικότητα. Υπάρχουν προβλήματα στα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει ένα μεγάλο κενό εφαρμογή όσον αφορά την ε, προστασία εθνοτικών, θρησκευτικών και ε, άλλων μειονοτήτων. Όσον αφορά τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους, ε, αντιμετωπίζονται με ατιμορρησία, ειδικά από την πλευρά κυβερνώντος κόμματος. Η Εκκλησία η Ορθόδοξη έχει συμμαχήσει με το κράτος και αυτό συμβάλλει στην ριζοσπαστικοποίηση της ε, κοινωνία ενάντια στις ε, μειονότητε, γιατί η κοινωνία της Γεωργίας τίνει πάντα να παίρνει το μέρος της Εκκλησίας. Αυτή είναι η γενική εικόνα σχετικά αφορά τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Υπήρξαν όμως δύο ε, υποθέσεις η μία έχει να κάνει τον, ε, τον Αφγάν Μουκτάρη, δημοσιογράφο του Αφγανιστάν, ο οποίο ε, απήχθη από άγνωστου ε, στη Τυφλίδα και μεταφέρθηκε στο Αζερβαϊτζάν. Εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών ε, θεώρησαν ότι αυτό έγινε με σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών ασφαλείας της Γεωργίας και της ε, αρχής του Αζερβαϊτζάν και μία άλλη υπόθεση αφορά έναν δάσκαλο τον ε, Μουστάφα Τσαμπούκ, ο οποίος ε, ε ανακρίθηκε και συνελήφθη τις ε, γεωργικές αρχές μετά από αίτημα των τουρκικών αρχών. Όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δέχτηκαν επιθέσεις και κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Σοκιασβίλη με δύο τρόπο η νέα κυβέρνηση άλλες μεθόδους για να μειώσει και να ελέγξει, να μειώσει την επιρροή τους και να τα ελέγξει. Χρησιμοποιεί εκβιασμούς των ιδιοκτητών των ε, τηλεοπτικών σταθμών που έχουν και άλλες επιχειρήσεις όπως είναι η περίπτωση του TVP Βέλη. Χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη, περίπτωση του Ρουστάβη 2 και με τη συγχώνευση καναλιών για να δημιουργήσει ένα κανάλι το οποίο θα είναι υπέρ της κυβέρνησης. Η Γεωργιανή Δημοκρατία αντιμετωπίσει προκλήσεις και από την Γεωργιανή Ορθόδοξη Εκκλησία. Παρόλο που είναι ένα κοσμικό κράτος, η Εκκλησία έχει αυξήσει την επιρροή της και στο κράτος και στην κοινωνία. Το κυβερνών κόμμα καθιστά την Εκκλησία ακόμα πιο ισχυρό παράγοντα και καλεί πολύ συχνά εκπροσώπους της Εκκλησίας στις συζητήσεις που γίνονται για την ομοθεσία. Έχω 30 δευτερόλεπτα. Έχουν, έχουμε και κάποιες θετικές εξελίξεις. όσον αφορά Όσον αφορά την νεολαία, έχουμε ε, πρόοδο στο θέμα με την ε, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολο Βέβαια, να είμαστε μέσα στο πλαίσιο της ανατολικής γειτονίας. Θα ολοκληρώσω εδώ. Θα μιλήσω για τις συστάσεις, αν θα σας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Και θα περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις. Πρώτη είναι η κυρία Κανιέτη. Ε, thank Σας ευχαριστώ και πάλι βάλτε τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω λετωνικά. Όσον αφορά τα δύο άλλα κράτη και όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Η δημοκρατία προφανώς λειτουργεί, αλλά αυτό που μας ανησυχεί είναι η κρατική διοίκηση που αναπτύσσεται παράλληλα με την αυστηρή στάση των κομμάτων Ιβανισβήλη. Έχει πολύ μεγάλη επιρροή στόχο τη γεωργία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορεί να προσχωρήσει κανεί αν το κράτο είναι κλεμμένο εισαγωγικά. Πρέπει να σκεφτούμε ότι μια πραγματική δημοκρατία λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί που έχουν την δύναμη, την εξουσία πρέπει να εκτιμούν και τη γνώμη της αντιπολίτευσης και να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το δικαστικό σύστημα. Κυρία Μούντι. Ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε για τη μελέτη σας. Τη διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον και θα συμφωνήσω με τα όσα είπε νωρίτερα ο κ. Στρεβίτσιος ότι ήταν πολύ καλή η πρωτοβουλία της Επιτροπής αυτής να ερευνήσει σε βάθος την εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης και το αποτέλεσμα των ε, σχέσεών μας, το πώς αναπτύσσεται στη χώρα δηλαδή, στις χώρες. Υπάρχουν ανησυχίες που εμείς έχουμε θέσει ως κοινοβούλιο στις ε, κυβερνήσεις. Την έλλειψη πρόοδου σε ορισμένους τομείς, ανησυχίες σε άλλους τομείς. Όμως, όταν διαβάζετε την εκθεσή σας, ε, όντως αναφέρεστε σε αυτές τις ανησυχίες, αλλά δεν υπάρχει αναγνώριση για κάποιες από τις αλλαγέ που έχουν λάβει η χώρα. Παραδείγματο χάρη αναφέρεστε στην εισαγγελία, αλλά δεν υπάρχει αναφορά στην εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στο διορισμό του επικεφαλής εισαγγελέα. Υπάρχει και αναγνώριση από την Transparency International ε, σχετικά. Και νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν καλό στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση της Γεωργίας έλαβε υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της Βενετίας και έκανε κάποιες αλλαγές και συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο. Σίγουρα η κυβέρνηση της Γεωργίας θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερα θετικά από όσα αναφέρονται στην εκθεσή σας. Και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να υπάρχει μεγαλύτερη αναγνώριση αυτών των στοιχείων. Ευχαριστώ πολύ. Γιούρεκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να σας ε, ζητήσω να αναφέρετε με περισσότερες λεπτομέρειες το ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Γεωργία. Αναφερθήκατε σε αυτό. Γιατί το γεγονό ότι η Εκκλησία είναι μέρος της κοινωνίας ε, είναι κάτι κανονικό. Έτσι λοιπόν υπάρχει η υποχρέωση να διεξάγεται ένας διάλογος ακόμη και με θρησκευτικές αρχές στις χώρες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, πιστεύετε ότι θα ήταν καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω οποιονδήποτε διάβλων, μέσω του πρεσβευτή μας στη Γεωργία ή μέσω άλλων διάβλων Πιστεύετε ότι θα ήταν καλή ιδέα να έχουμε έναν πιο βαθύ διάλογο με σημαντικούς θρησκευτικού θεσμούς ε, στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Γιατί αν αυτές οι θρησκευτικές αρχές πιστεύουν ότι αγνοείται η δική τους άποψη, τότε θα διατυμπανίσουν τις απόψεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια υποχρέωση που θα πρέπει ίσως να επιβληθεί από τα κρατή-μέλη στους ε, ευρωπαϊκούς, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τι πιστεύετε λοιπόν ε, για το διάλογο μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχω το ίδιο σχόλιο ε, για την Ουκρανία. Όταν θα συζητήσουμε για την Ουκρανία θέλω να θέσω την ίδια ερώτηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στετίνα. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω τσεχικά. Βάλτε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, κύριε Μιχελίτσα. Μας παρουσίασατε δύο κυρία σημεία πολύ ξεκάθαρα σήμερα. Μας είπατε ότι ε, υπάρχει πρόοδος στη Γεωργία, αλλά μας είπατε ότι υπάρχουν και πολιτικοί κρατούμενοι στη Γεωργία. Δηλαδή, τι εννοούσατε ότι αφού ανέλαβε την εξουσία το Γεωργιανό όνειρο, υπήρξε μία έρευνα κατά μελών της προηγούμενης κυβέρνησης ε, και 30 από αυτούς καταδικάστηκαν, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος σας Καρβίλη. Αυτό εννοούσατε. Γιατί πολύ συχνά συζητάμε για το ότι η Γεωργία έχει επιλεκτική δικαιοσύνη. Αυτό εννοούσατε. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γκάλερ. Yes, uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Συνολικά θα λέγατε ότι πηγαίνουν προς θετική κατεύθυνση. Δεν θέλω να συγκρίνω ως ίσο προς ίσο τον κύριο Βενισβίλη με τον κύριο Πλατχόνιουκ ε, στο πώς χειρίζονται τα πράγματα. Όμως, από δομική σκοπιά είναι αυτή που είναι ουσιαστικά στα παρασκήνια. Και υπάρχει ένας παραλληλισμός του κυρίου Βενσφίλ με την κατάσταση στη Μολδαβία. Αλλά δεν θα ήθελα να μπω σε σύγκριση σε σχέση με την πολιτική που ασκείται. Σίγουρα η κατάσταση στη Γεωργία είναι πολύ καλύτερη και σταθερή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Σύνταγμα εσείς ε, θα θεωρήσετε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος ε, στον τομέα αυτό, όταν φυσικά θα εφαρμοστεί ε, κατά γράμμα και κατά πνεύμα. Είδαμε και την αξιολόγηση της Επιτροπής της Βενετίας και υπήρξε κάποια αλληλεπίδραση. Υπήρξε αντίδραση, εξετάστηκαν αποκλίνουσες απόψεις σε σχέση με το αρχικό κείμενο με το αρχικό σχέδιο κειμένου. Γενικά θεωρούσα ότι αυτές είναι θετικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σόνιετς ως τελευταίος ομιλητής. Θα ήθελα κι εγώ να ρωτήσω για τους εκπρόσωπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας ε, της Γεωργίας, ε, κυρία Μιχελίτσε. Εσείς αναφερθήκατε σε αυτό σαν να είναι λάθος να συναμιλούμε με τα μέλη των θρησκευτικών οργανώσεων στην Ευρώπη. Όμως, ε, το χάρη, ε, γιατί είναι καλύτερο να συνομιλούμε παραδείγματος χάρη με ανθρώπους που εκπροσωπούν ε, ε οργανώσεις ομοφιλοφίλων παρά με εκπροσώπους θρησκευτικών ε, οργανώσεων Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, ε, κάποιο αποκλείστηκε από την Κομισιόν επειδή θεωρήθηκε ότι είναι πιστός καθολικός. Έτσι, λοιπόν, είναι υποκριτικό απλώ ε, απλώς κατ' επίφαση να δηλώνουμε ότι είμαστε ουδέτεροι, γιατί ρητορική μίσους είναι ένας όρος, παραδείγματος χάρη μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ε, αν κάποιος πει ότι η ομοφιλοφιλία ε, είναι Είναι μια εκτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε πέντε λεπτά για να απαντήσετε αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις. Ε, ναι, είναι κάπως δύσκολο να απαντήσω. Γιατί είχαμε κάποιες ε, παρόμοιες ερωτήσεις επίσης. Λοιπόν, δημοκρατία και σεβασμό ε, για την πολυτελήτευση. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για τη Γεωργία ήταν ε, μεγάλη πρόκληση από την ανεξαρτησία γιατί έχουμε τη λογική ο νικητή παίρνει τα πάντα. Σε περιφερειακό, τοπικό επίπεδο, εθνικό επίπεδο. Και εδώ φτάνουμε στους πολιτικούς κρατούμενους. Ναι, αναφέρθηκα σε αυτούς που είναι ε, φυλακισμένοι και είναι μέλη της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτούς. Όταν ε, μίλησα για πολιτικούς κρατουμένους, ε, για αποφάσεις που είναι πολιτικά, που είναι δυνάμει πολιτικής επιρροής, αναφέρθηκα και σε αποφάσεις που αφορούν δημοσίους επιλήλους όσοι θεωρήθηκαν ότι υποστήριζαν την προηγούμενη κυβέρνηση έχουν απολυθεί από διάφορα τμήματα, από υπουργεία ή από τους δήμους. Αυτό εννοούσα υπό την επιλεκτική δικαιοσύνη. Και φυσικά συμφωνώ με τις θετικές εξελίξεις. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, ήταν ε, ίσω αρκετά θετική απέναντι στη Γεωργία, όμω αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να αποτρέψουμε να, να καταλήξουμε στην κατάσταση τη Μολδαβία. Νομίζω καλύτερη είναι πρόληψη παρά να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, τι συνέπειε. Σίγουρα είναι μια ιστορία επιτυχία η Γεωργία, αλλά εντό του πλαισίου τι ε, εταιρικέ σχέσει έχουμε τον Λουκασένκο, έχουμε και τον Άλεφ. Ε, έτσι λοιπόν είναι πολύ εύκολο σε αυτό το πλαίσιο να αποτελεί κανεί ιστορία επιτυχία. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα. Ποιε είναι οι προσδοκίε του πληθυσμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει και σύγχυση με την προοπτική ένταξης. Φαίνεται σαν η Ευρωπαϊκή Ένωση να επενεί τη Γεωργία για την ανάπτυξη των κρυκοθεσμών και αναρωτιέται ο κόσμος γιατί αφού είμαστε τόσο καλοί ε, δεν μας δίνει την προοπτική ένταξη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αρχίζουν να μιλάνε για την Ρωσία, για την πολιτική της Ρωσίας, ένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Θα πρέπει να είστε αρκετά και να πείτε ότι ξέρετε δεν σας δίνουμε την προοπτική ένταξη γιατί έχετε πραγματικά προβλήματα ε, ως προς την ανάπτυξη της δημοκρατίας. Και συμφωνώ μαζί σας, υπάρχουν ε, θετικές εξελίξεις, υπάρχει πρόοδος στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Η χώρα επιτυχώς καταπολέμησε την διαφθορά σε χαμηλά και σε μεσαία επίπεδα, αλλά στη συνέχεια έχουμε τη διαφθορά στην ελίτ. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το μετρήσει η Transparency International, γιατί η μεθοδολογία ε, που χρησιμοποιεί βασίζεται στην αντίληψη του πληθυσμού. Και φυσικά ο πληθυσμό συνήθω δεν ε, έχει την ενημέρωση για τη διαφθορά σε υψηλά επίπεδα, γιατί μιλάμε για συμφωνίες που γίνονται μεταξύ των πολιτικών, μεταξύ των πολιτικών και των επιχειρηματιών. Συνήθως λοιπόν ε, τα αποτελέσματα αποτελέσματα αυτά δεν καταλήγουν στις εκθέσεις της Transparency International. Τώρα για την Ορθόδοξη Εκκλησία βεβαίως είναι σημαντικός παράγοντας στη χώρα και φυσικά ο διάλογος είναι πάντοτε κάτι θετικό. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει αρχίσει να συνομιλεί με την Ορθόδοξη Εκκλησία και ξέρω ότι πρόσωπος ε, της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχει επισκεφτεί τις Βρυξέλλες ε, και ήταν πολύ ικανοποιημένοι γι' αυτό και ίσως κάποιος να άλλαξε, από αυτούς να άλλαξε γνώμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως, ε, ως θεσμό και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένταξη όμως το πρόβλημα που εντοπίζω είναι το εξής. Υπήρχε ένα παράδειγμα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να νομοποιήσει κάποιες ε, κατηγορίες σε πολιτική διαδικασία. Παραδείγματο χάρη υπήρχε μία ε, συζήτηση που αφορούσε την νομοθεσία κατά της διαφθοράς. Ε, και η Εκκλησία ήταν κατά ε, επειδή ε, δεν θέλει να θεωρείται διάκριση, διάκριση που γίνεται βάσει θυσίου προσανατολισμού. Έτσι λοιπόν νομοποιούνται κάποιες δημοσκοπήσεις σε αυτό το θέμα και τελικά έμεσα συνεισφέρει στη ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας, γιατί στις περιπτώσεις αυτές η κοινωνία συνήθως η πάντα τίνει να ακολουθεί την άποψη της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα περάσουμε στην τρίτη μελέτη για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ουκρανία. Έχετε 10 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ εξότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ που με καλέσατε να συμμετάσχω σε αυτήν την ε, συλλογική ε, προσπάθεια για την αποτίμηση της προόδου σε ό,τι αφορά τις ε, συμφωνίες σύνδεσης και πιο συγκεκριμένα αυτή για την Ουκρανία. θα διαβάσω το κείμενό μου γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να μείνω στο δεκάλεπτο και ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα να πω το προφανές, το οποίο όμως δεν είναι μελιτέο. Όταν εξετάζουμε την ε, πρόοδο σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, αλλά και τις προκλήσεις για την Ουκρανία. Η Ουκρανία λοιπόν ε, βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση και στο εσωτερικό της για την μεταπαραθετική σταθεροποίησή της και με βάση τις αυξανόμενες εξωτερικές πιέσεις οι οποίες εντείνονται και από την ρωσική προσάρτηση της Κρυμαίας αλλά και ε, για την επιθετικότητα της Ρωσίας στον Βάσ αλλά και τις ε, πρακτικές της Ρωσίας στην θάλασσα του Αζόφ. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης και το φιλόδοξο ε, ε, θεματολόγιο μεταρρυθμίσεων για αυτή τη χώρα τίθεται ένα αμφιβόλο από μια ε, μεγάλη γκάμα αρνητικών κοινωνικοπολιτικών, οικονομικών και νομικών παραγόντων. Ωστόσο, σημαντική προοδο έχει σημειωθεί σε πολλου τομει ομω παραμένει η πρόκληση να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση σε τομείς που μέχρι τώρα έχουν μείνει πίσω. Και το πιο σημαντικό είναι να συνεχιστεί η διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Θα σταθώ σε τέσσερις ε, πυλώνες. Το θεσμικό ε, πλαίσιο, νομική και ε, ρυθμιστική προσέγγιση, υλοποίηση ε, της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών και οι μεταρρυθμίσεις για κυβέρνηση στην Ουκρανία. Το πρώτο λοιπόν, θεσμικό πλαίσιο. Η υλοποίηση της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ άλλων και με την μεταφορά στο δίκαιο της Ουκρανίας ενός ε, μεγάλου τμήματος ενωσιακής νομοθεσίας με 564 ε, νομικές πράξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια πολύ σημαντική θεσμική πρόκληση. Σε ό,τι αφορά τώρα το θεσμικό πλαίσιο τη διαδικασία υλοποίησης, η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ουκρανία δεν είναι πλέον το επίσημο μοντέλο συντονισμού το οποίο πλέον εποπτεύεται από ε, το σχετικό, τον αρμόδιο φορέα, ε, αλλά πλέον τίθεται το ζήτημα της ε, θεσμικής και διοικητικής ικανότητας των δημοσίων αρχών να ελοποιήσουν τη Συμφωνία Σύνδεσης. Και αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, γιατί είναι αναπολετασματική η δημόσια διοίκηση της Ουκρανίας. Τον Απρίλιο του 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ξεκίνησε το project EU4PAR στην Ουκρανία. Ένα τετραετές ε, πρόγραμμα ε, με στόχο μια πιο αποτελεσματική και υπεύθυνη δημόσια διοίκηση. Από τον Αύγουστο η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε 15,5 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Η αύξηση της οικονομικής βοήθειας είναι αποτέλεσμα της προόδου που έχει σημειωθεί με τις μεταρρυθμίσεις. Σε μία ε, μελέτη που δημοσιοποιήθηκε το 2018 αναφέρθηκε ε, και, και από το πρόγραμμα ΣΥΓΜΑ ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος ό,τι αφορά τη δημόσια διοίκηση. Όμως υπάρχει ανισομέρεια ε, σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ε, τα πηγαίνει καλύτερα σε σχέση με άλλους τομείς. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ε, ε, προσέγγιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Έχουμε λοιπόν χαμηλούς ρυθμούς προσέγγισης και καθυστερήσεις στη μετάφραση του ευρωπαϊκού κεκτημένου στην Ουκρανική. Το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας και της υλοποίησης της συμφωνίας χαρακτηρίζεται και από μία ε, όχι τόσο ιδανική ε, απόδοση των ε, κρατικών θεσμών και χαμηλό, υπάρχει χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνη από την Ουκρανική κοινωνία. Αυτή η χαμηλή εμπιστοσύνη επηρεάζει και την στήριξη που υπάρχει προς ε, συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, ιδίως σε κάποιες που δεν είναι δημοφιλείς. Περνάω τώρα στο δεύτερο άξονα, νομοθετική προσέγγιση και εφαρμογή του νόμου. Εδώ υπάρχει καλός ρυθμός, αν και θα μπορούσε να είναι καλύτερος. Είναι όμως δύσκολη η διαδικασία υλοποίησης. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες στην υλοποίηση εντοπίζονται σε δύο τομείς. Τεχνικά προσκόμματα στο εμπόριο, σε ό,τι αφορά την νομοθεσία πλαίσιο και ενεργειακή απόδοση των κτηρίων που οφείλεται και στο υψηλό ε, επίπεδο ενδιαφέροντος ε, και συμμετοχής και των εσωτερικών ε, ενδιαφερομένων μερών. Ο δεύτερος τομέας είναι ο τομέας των ε, δημοσίων ε, προμηθειών και διαγωνισμών. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα τομείς ε, που αποτελούν προόκληση, φορολογία, τελωνία, εταιρικό δίκαιο και προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Ιδίω σε ό,τι αφορά τα τελωνία υπάρχει υψηλή διαφθορά με τεράστια ε, διαρροή κεφαλαίων και απώλεια κερδών από αυτή την άποψη. Η Süddeutsche Zeitung αναφέρει ότι περίπου 5 δις ευρώ ε, είναι οι δημοσιονομικές απώλειες της Ουκρανίας εξαιτίας των, της διαφθοράς στις θελωνιακές επιχειρήσεις. Δύο Τώρα για την ε, εφαρμογή της ε, σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθερών συναλλαγών. Το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2016 μέχρι σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον είναι ο υπαριθμόν ένα εμπορικός εταίρος ε, της Ουκρανίας και έχει, έχει αντικαταστήσει τη Ρωσία. Με αυτή την εξέλιξη λοιπόν υπάρχει μία αύξηση ε, του ΑΕΠ κατά 2%. Τα τελευταία χρόνια η Ουκρανική οικονομία και έχει σταθεροποιηθεί, αλλά έχει δείξει και σημάδια βελτίωσης. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2017. Οι εξαγωγέ της Ουκρανία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 30,4% και έφτασαν ε, σε επίπεδα ρεκόρ των 17,5 δι δολαρίων που είναι το ανώτατο σημείο από το 2012. Η αύξηση των εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχει άμεσο αντίκτυπο και στην χρήση ή και εξάντληση των ε, ποσοστώσεων ε, δασμολογικών συντελεστών, TRQs και έτσι πρέπει να ενταθεί ο διάλογος για την προσαρμογή και τροποποίηση αυτών των συντελεστών. Τέταρτον τώρα, μεταρρυθμίσει ε, χρηστή διακυβέρνηση. Υπάρχουν σημαντικέ μεταρρυθμίσει, αλλά δεν προχωρούν όλε ε, με σταθερό ρυθμό. Το μοναδικό παράδειγμα ε, που πλέον έχει ολοκληρωθεί είναι η αποκέντρωση. Κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις, όπως αυτή κατά της διαφθοράς ε, και στον τομέα της δικαιοσύνης, μπορεί να σταματήσουν την πορεία τους μετά από τις ε, εκλογές του 2019. Η εξωτερική θεσμική και πολιτική στήριξη είναι εξαιρετικά σημαντική εδώ, ε, καθώς παραδοσιακά η εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τις δημόσιες αρχές είναι πολύ χαμηλή. Τέλος, να μιλήσω για την αναγκαιότητα της παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η υλοποίηση ε, της Συμφωνίας Σύνδεσης ε, δέχτηκε πολλές πιέσεις από αρνητικές οικονομικές, κοινωνικοπολιτικές και άλλες εξελίξεις. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε λοιπόν αυτούς τους παράγοντες και αυτές τις εξελίξεις όταν εξετάζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί χρειαζόμαστε μια ρεαλιστική προσέγγιση που θα ιεραρχεί προτεραιότητες τη φορά την πρόοδο που σημειώνεται στην Ουκρανία. Μέχρι τώρα είναι υπερφιλόδοξες ε, οι εκτιμήσεις και από τις δύο πλευρές. Πρέπει λοιπόν να είναι βιώσιμη η διαδικασία μεταρρυθμίσεων και μη αντιστρέψιμη. Αυτό θα πρέπει να είναι το βασικό μέλημα Βρυξελών και Κιέβου για το επόμενο 1,5 έτος. Υπάρχει ε, σημαντική λαϊκή βούληση για μια τέτοια πολιτική εξέλιξη. Με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις του Αυγούστου, 66% των Ουκρανών εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 70% του πληθυσμού θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ένας τρόπος βελτίωσης της πολιτικής σταθερότητας και ασφάλειας στη χώρα. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους σας ευχαριστώ και με στη διάθεσή για ερωτήσεις. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκάλερ καταρχήν. Yes, uh, thank you very much uh, for this uh, overview. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επισκόπηση. Θα έλεγα ότι συμφωνώ με τα πορίσματά σας σε μεγάλο βαθμό. Σε σχέση τώρα με την ικανότητα να αντιμετωπιστούν παράλληλα όλες οι μεγάλες προκλήσεις πού θα συνιστούσατε να γίνει ο κύριος συντονισμός. Δηλαδή βλέπω ότι έχουμε συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, όμως δεν υπάρχει συντονισμός και δεν υπάρχει πολλή επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων. Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση. Εσείς ε, πού θα εντοπίζετε την ανάγκη του συντονισμού, θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο πρωθυπουργού, σε επίπεδο προέδρου, αυτές είναι ίσως οι κύριες επιλογές στη δημοσία διοίκηση και για τα τελωνία. Αναφερθήκατε στο άρθρο της ε, γερμανικής εφημερίδας, το διάβασα και εγώ. Όμως, ναι, όντως, χάνεται ένα πολύ μεγάλο εισόδημα. Με μεγάλη πηγή εισοδήματο. Γιατί κάποιοι ε, αρπάζουν τα χρήματα του κράτους. Ποιοι είναι αυτοί. Έχετε φτάσει τόσο εις βάθος ώστε να τους προσδιορίσετε, να τους εντοπίσετε. Πρόκειται για συντονισμένες ε, δράσεις Ποιος κάνει τι, πώς λειτουργεί όλο αυτό και πώς ε, ουσιαστικά συμβαίνει αυτό εφόσον όλοι γνωρίζουν ότι αυτά συμβαίνουν στον τελωνιακό κλάδο και πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καλνιέτ. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Μάικλ Γκάλ. Θα μιλήσω όμως στα λιτωνικά. Φορέστε τα ακουστικά σας. Η Ουκρανία είναι ένα κράτος υποκατοχή. Συνεχίζει ο πόλεμος, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για την πολιτική εξουσία Η διαφθορά λειτουργεί βάρος των συμφερόντων. Κανείς δεν διαμαρτύρεται ενάντια σε αυτό. Είναι σωστά αυτά που τονίζεται στην έκθεση ότι το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφοράς είναι ανεπαρκές. Πολλά ελέγχονται από τους ολιγάρχες. Το δικαϊκό σύστημα δεν είναι αποδοτικό, αποτελεσματικό. Γι' αυτό θεωρώ ότι καθήκον μου είναι να προειδοποιήσω ότι η υπομονή του Ουκρανικού λαού δεν είναι ανεξάντλητη. 70% των Ουκρανών εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, και, ότι η κυβέρνηση μπορεί να έχει την ίδια εμπιστοσύνη. Είναι ιστορικά υπεύθυνη με στι εκλογέ η κυβέρνηση και πρέπει να διαχειριστεί τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ώστε το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών είναι τέτοιο. Ο λαός να πιστέψει ότι δεν θα επικρατήσει χάος και αυτό μπορεί να αλλάξει χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τέλος της καριέρας μου, με τον Brexit να πλησιάζει ως πολιτικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμάμαι το γεγονός ότι είχα γράψει ένα άρθρο στο 2002 λέγοντας ότι η Ουκρανία έχει προοπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι ότι μετά από μια δεκαετία, παραπάνω από μια δεκαετία, Κροατία, 70% του λαού συμφωνεί μαζί μου και εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιθυμούν να το δουν αυτό ως μέλλον. Είναι καλό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δικαστεί στη Ρωσία ως βασικό εμπορικό εταίρο. Υποστηρίζω αυτή την πρωτοβουλία να μιλήσουμε για τις τρεις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Η Ουκρανία είναι η πιο σημαντική λόγω του μεγέθους της και την επιρροή της στον κόσμο. Και βρίσκεται ακόμα φυσικά υπό μεγάλη οικονομική και πολιτική πίεση με την ε, κατοχή στην Κρυμαία και την ε, διαμάχη που συνεχίζεται. Η ερώτησή μου, στατιστική 1 προς 5 για τα τελωνία και για τη διαφθορά και τους ολιγάρχες που είχα να κάνουν με τις ε, τελωνιακές αρχές. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με δύο σημεία στην έκθεση. Την ανάγκη να υπάρξει από ολιγαρχοποίηση στην δυτικοποίηση κάποιων φορέων και όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά πόσο η κυρία κύριος Τούσκα βλέπει ότι η ίδρυση ενός ε, δικαστηρίου ενάντια της διαφθοράς που θα αντικαταστήσει το αρμόδιο γραφείο το οποίο πράττει έκανε εξαιρετικό έργο Ποια θα είναι, θα είναι του δικαστηρίου, γιατί η διαφθορά είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για την ε, ανισορροπία στην διάθεση των πόρων. Ο κύριο Τάνο και ο κύριο Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους συμπυρογνώμονες στην ομάδα. Εξαιρετική η μελέτη που μπορεί να φανεί χρήσιμη σε πολλούς πολιτικούς και αυτούς που έχουν ε, να κάνουν, να με τις μεταρρυθμίσεις. Θα θέλαμε να έχουμε τη μετάφραση και στα Ουκρανικά, όπως και στα Ρουμανικά και στα Γεωργιανά αντίστοιχα τις άλλες μελέτες. Έχετε κάποια συγκεκριμένη άποψη για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ε, στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πολλά όσον αφορά την τομεακή στήριξη. Έχουμε μια ομάδα με επιφαλή στον Πίτερ Βάγνερ καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες, αλλά βλέποντας τελικά αποτελέσματα κατά ποια είναι τα αποτελέσματα που αναμένουμε να έχουμε. Και το δεύτερο, υπήρξε μια αρισμότητα για την Ουκρανία όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διάρκεια του 2017 υπήρξε ένας διάλογος με τις Ουκρανικές αρχές που που οδήγησε σε αναστολή της ε, μακροοικονομικής ε, ενίσχυσης. Πώς το εξέλαβαν αυτό οι πολιτικές ελίτ στην Ουκρανία και πώς το κοινό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταίος συνάδελφος, ο κύριος Σαφχάουσερ. Μάλιστα, θα ήθελα ε, και εγώ να πω κάτι για, τους, ε, για τα τρία αυτά ζητήματα των τριών χωρών. Αρχικά πρόκειται για τρία αποτυχημένα κράτη. Ε, έχουν περιοχές ε, με αποσχεστικές τάσεις και οι τρεις χώρες και ως αιτία Κρυμαία, Ντονμπάς και το καθεξής. Τρία λοιπόν αποτυχημένα κράτη λοιπόν. Ε, με ιστορική σχέση και εξάρτηση από τη Ρωσία. Οπότε πάντα υπάρχει μια διελκυστίνδα μεταξύ των φιλοευρωπαϊκών και φιλορωσικών τάσεων. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, ε, τρία διεφθαρμένα κράτη. Για τη Μολδαβία είναι ξεκάθαρα με το ένα δις που εξαφανίζεται. Και για την Ουκρανία τώρα αναφέρθηκε προηγουμένως για τα πέντε δις Υπάρχουν πολλά δισεκατομμύρια που εξαφανίζονται ω διαμαγεία. και ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει ελαφρά την καρδία να ε, υποστηρίζει και να τροφοδοτεί αυτά τα μαφιόζικα δίκτυα. Τρία αποτυχημένα κράτη, τρία διεφθαρμένα κράτη. Επόμενη διαπίστωση. Αυτή η ηθικοπλαστική προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης έχει φτάσει στο τέλος της. Όταν ε, βλέπουμε τις απτές προεκτάσεις της πολιτικής μας ε, και στην Ουκρανία και στη Μολδαβία. Στην Ουκρανία όπου στηρίζουμε τους ε, διαρρευθυνμένους πολιτικούς. Ε, στη Μολδαβία τώρα λέμε ότι α, ίσως δεν θα έπρεπε να είχαμε υποστηρίξει αυτό τον πλήρως διεφθαρμένο φιλοευρωπαϊστή, καθώς έχουμε έναν φίλο Ρώσο πρόεδρο. Στην Ουκρανία συνεχίζουμε όμως να δίνουμε χρήματα σε διεφθαρμένους και μάλιστα χρήματα που εξαφανίζονται. Επόμενη διαπίστωση. Πλήρη ασυνέπεια στην πολιτική μας. Στον Τον μιλούμε για στρατιωτική επίθεση και προσάρτηση. Πολύ καλά. Βέβαια, αυτό αντιτίθεται στις ε, συμφωνίες του Μίνσκ. Έχουμε λοιπόν μια πολιτική που αντιτίθεται στις συμφωνίες του Μίνσκ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά για τη Γεωργία διακόπτει ο πρόεδρος ε, και στην ε, Μολδαβία Είμαστε κατά του δημοψηφίσματος που όμως είχε 90% υποστήριξη για την τρανσδινιστερία. Και όλα αυτά επειδή δεν υπάρχει κλίνο, Πρόεδρε, γιατί δεν υπάρχει ε, γεωπολιτική προσέγγιση. που, δεν θέλει να διχάσει την Ευρώπη, αλλά θέλει να τη ε, συγκεράσει και τη Δύση και την Ανατολή. Ευχαριστούμε. Περνάμε στι απαντήσει για πέντε λεπτά. Ε, Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ανησυχώ πώς θα τις απαντήσω όλες επαρκώς. Στο χρόνο που μου δίνετε, αλλά θα ξεκινήσω με τη σειρά που τις θέσατε. Πρώτον, Ευχαριστώ τον κύριο Γκάλερ που μοίρασε τα αποτελέσματα της ε, έκθεσης και ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Η βασική ανησυχία για το που θα πρέπει να εστιάσει η προσπάθεια συντονισμού απαντήσετε μόνο σας, θα πρέπει να είναι ο Πρωθυπουργός και το αρμόδιο γραφείο για την ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ αναγνωρίζω. Στον πληθυσμό ότι είναι υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία στην Ουκρανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κυβέρνησή μας ξεκίνησε μια ε, εκστρατεία ενημέρωσης όχι μόνο για να ενημερώσει τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ένωσης ε, στην Ουκρανία γιατί 70% των Ουκρανών δεν γνωρίζανε για την ενίσχυση που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ουκρανία ούτε για τα προγράμματα δεν είναι ενημερωμένοι που λαμβάνουν χώρα. Παράλληλα αυτό είναι μια προσπάθεια να αλλάξουμε τον πολιτικό κύκλο στην Ουκρανία συμπεριλαμβάνοντας την, ε, ε, την ενημέρωση προς δύο κατευθύνσεις προς τον πληθυσμό σχετικά με την νομοθεσία, αλλά να ενημερώνουμε παράλληλα και για τα αποτελέσματα, για την επίδραση που θα έχει η νομοθεσία στον πληθυσμό. Αυτές είναι οι δύο βασικές αποστολές, τις οποίες ε, τις ε, προωθούμε σε συνεργασία με την Αντιπροσπέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το αρμόδιο κυβερνητικό γραφείο. Όσον αφορά την επόλυα πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Είναι δύσκολο να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση. Πώς αξιολογείται αυτή η απώλεια, οι στατιστικές από το Eurostat. Ε, μελετάνε πώς εισάγονται στην Ουκρανία, ενώ από την πλευρά της Ουκρανίας ε, αυτό που ε, μελετούν είναι πόσοι, πόσοι φόροι καταβάλλονται και αυτό που, παρα, 5 εκατομμύρια Ενδεχομένως λοιπόν θα χρειαστεί να δούμε το θέμα πιο εμπεριστατωμένα. Το δεύτερο ερώτημα που αφορά τα διλήμματα που αντιμετωπίζουμε αυτή την ώρα. Από τη μία πλευρά έχουμε την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ε, δικαιοσύνη για όλους και από την άλλη πλευρά, τουλάχιστον αυτό παρατηρούμε, τις προσπάθειες του καθεστώτος να αυτοσυντηρηθεί κάτι που είναι λογικό για οποιοδήποτε καθεστώς. Και αυτό είναι και εμφανές από την εμπιστοσύνη που έχει ο λαός στον πρόεδρο 20% του λαού εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Οι καθυστερήσει στη δημιουργία του ανώτου δικαστηρίου εναντί στη διαφθορά όταν θα ξεκινήσει τη λειτουργία του θα ε, επιχειρήσει να αντιμετωπίσει δύο διαμετρικά αντίθετα θεματολόγια ταυτόχρονα. Ένα άλλο ερώτημα για το μέλλον, το ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας. Ο πληθυσμός είναι φιλοευρωπαϊκός και αυτό αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στις ε, τελευταίες καταμετρήσεις, αλλά και τις προσπάθειες ε, που έγιναν ε, με τις τρεις επαναστάσεις. Γίνεται προσπάθεια να υπάρξουν τα συνταγματικά πλαίσια γιατί οι προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή και στο ΝΑΤΟ θεωρούνται ε, επιθυμητά και ο λαός δεν ήθελε να ξέρει ότι αυτό, αυτή η προοπτική δεν, θα τους αφαιρεθεί, δεν θα τους στερηθεί στις επόμενες εκλογές. Ο βουλευτής από το Ινωμένο Βασίλειο ρώτησε για την ε, καταπολέμηση της διαφθοράς και τι συμβαίνει εκεί. Πολλοί πυρογνώμονες θεωρούν ότι το δικαστήριο θα ξεκινήσει τις λειτουργίες του το τέλος του χρόνου, άλλοι λένε ότι δεν θα συμβεί μέχρι τις επόμενες εκλογές το 2019. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η διαδικασία ε, συνεχίζεται με την επιλογή ε, δικαστών, υποψηφιότητες που βουλήθηκαν τον Αύγουστο, στις 15 Σεπτεμβρίου τα διαφερόμενα ε, μέρη από άλλες χώρες θα έρθουν να κάνουν τις προτάσεις τους. για να αποφασίσουν για την τελική σύσταση του δικαστηρίου και προφανώς οι 600 εκκρεμείς υποθέσεις που διαχειρίζεται το γραφείο ενάντια στη διαφθορά δεν θα μπορούσαν να επιληθούν άμεσα. Θα σας ενθαρρύνω να δείτε καλύτερα το έγγραφο το οποίο έχει περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή της ε, συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ στους τρεις ε, Ευχαριστώ πολύ και τους τρεις ε, ομιλητές. Ε, σας ακούσαμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο. Continuamos, ¿no? Continuamos. Θα εξετάσουμε τώρα το σχέδιο έκθεση που έχει εκπονήσει ο συνάδελφο Αστροβίτσιο σχετικά με την εφαρμογή τη Συμφωνία Σύνδεση τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Μολδαβία. Να πω ότι μας ανησυχούν ιδιαίτερα τα νέα που φτάνουν από τη Μολδαβία. Υιοθετήθηκε τον περασμένο μήνα ένα έκτακτο ψήφισμα στο Στρασβούργο και επίσης ε, ε, υπήρξε και μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μπορώ να πω ότι δεν βλέπουμε σημαντική πρόοδο για τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις ε, στην Μολδαβία, λαμβάνοντας υπόψη ότι πλησιάζουν και οι βουλευτικές εκλογές. Χωρίς χρονοτρεβή θα δώσω το λόγο στον κύριο Αουστρεβίτσιους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ικανοποίησή μου να σας παρουσιάσω το σχέδιο της έκθεσης ε, για την Μολδαβία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τη Συμφωνία Σύνδεση ε, τέσσερα χρόνια μετά την υπογραφή τη Συμφωνία Σύνδεση από τη Μολδαβία και δεσμεύτηκε να προβεί σε οικονομικές ε, και πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Τα σημερινά πορίσματα παρουσιάζουν μια αντιφατική εικόνα της εφαρμογής ε, της συμφωνία σύνδεση. Ουσιαστικά είδαμε κάποιες θετικές εξελίξεις σε κάποιους τομείς, όπως ε, στον χρηματοπιστωτικό και τον τραπεζικό τομέα, σημαντική αύξηση στο διμερές εμπόριο και καλύτερο κανονισμό για τις επιχειρήσεις, καλύτερος κανονισμός από τις επιχειρήσεις. Όμως υπάρχουν εξελίξεις που έχουν επισκιαστεί από τη συνεχή επιστοδρόμηση των ε, πολιτικών και δημοκρατικών προτύπων, ε, το κράτος δικαίου και η ελευθεροτυπία και οι ε, κατάστασεις κοινωνίας των πολιτών είναι απογοητευτικές. Η έκθεση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μόλις μας παρουσιάστηκε μας ε, δείχνει ότι το συνολικό αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκε στη Μολδαβία θα πρέπει να θεωρηθεί ως μη ικανοποιητικό. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μολδαβία συνεχίζουν να είναι στενοί εταίροι, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε ποιους τομείς ε, περιμένουμε διαφορετικό ρυθμό μεταρρυθμίσεων και δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τα σημερινά επιτέγματα. Πέρσι, ε, ο ε, νόμος, η αλλαγή του εκλογικού νόμου που δέχτηκε κριτική, από την Επιτροπή της Βενετίας εξακολουθεί να παραμένει εμπόδιο για διαφανείς εκλογικές και δίκαιες εκλογικές διαδικασίες. Η μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος, η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, το κράτος δικαίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει να συνεχιστούν και να επιταχυνθούν. Γι' αυτό η πρόσφατη απόφαση να απομακρυνθεί ο Ντορίν Κερτοάκα από τη Δημαρχία του Κισινάου και να ε, κληρωθεί η εκλογή του Αντρέινα Στάση παραμένουν σοβαρή ανησυχία για πολλά θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να ανησυχεί για σημάδια περαιτέρω συρρήκνωση ε, τη κοινωνία των πολιτών στη Μολδαβία. Επιπρόσθετα, το πρόσφατο δέσμη μέτρων για τη φορολογική μεταρρύθμιση, για την αμνηστία του κεφαλαίου και για φορολογικά κίνητρα θα πρέπει να αναλυθεί πλήρω, καθώ μπορεί να περιορίζει την ικανότητα της Μολδαβίας να καταπολεμήσει τη διαφθορά και την ομιμοποίηση παράνομων εισόδων. Λαχθόντων αυτών, Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει την αρχή της αιρεσιμότητας στην μακροοικονομική βοήθεια και οποιαδήποτε μελλοντική ε, μακροοικονομική βοήθεια θα πρέπει να δοθεί αφού έχουν οριστεί οι εκλογές του Φεβρουαρίου 2019 θα πρέπει ουσιαστικά να γίνουν σεβαστά τα διεθνή πρότυπα. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να συνεχίσουμε το σημαντικό μας διάλογο με τις αρχές και την κοινωνία των πολιτών της Μολδαβίας. Αυτό προκειμένου να εγγυηθούμε πλήρη κατανόηση και τιμότητα για μελλοντική συνεργασία, που περιμένω να είναι πιο αποτελεσματική και πιο εξορθολογισμένη για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τον συνάδελφο Ζουλιάν ε, για τη μεγάλη υποστήριξη στην υλοποίηση της έκθεσης. Ανυπομονώ να λάβω τα σχόλια, τις τροπολογίες και τις προτάσεις σας ε, για την κατάρτιση του τελικού κειμένου. Επίσης, θα ήθελα να έχουμε περαιτέρω συζητήσεις για τη Μολδαβία, καθώς Μόνο αν συνεχίσουμε να είμαστε εταίροι με τη Μολδαβία μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία σύνδεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αστροβίτσιο. Να δώσουμε το λόγο στους προσκεκλημένους από την Κομισιόν. Το αντίθετο μου λένε, όχι. Πρώτα θα ακούσουμε τους βουλευτές. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ. Θέλω να διαβάσω κάτι εκ μέρου του κ. Κόβατσεφ που είναι σχέδιο συζητητής και ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Παραθέτω. Θα ήθελα να ευχαριστήσει τον εισηγητή για τη σκληρή δουλειά επί της έκθεσης αυτής που παρουσιάζει τα κυρία σημεία ανησυχία για την εφαρμογή της Συμφωνίας σύνδεση με τη Μολδαβία έτσι όπως έχει εκφραστεί πολλές φορές ενώπιον αυτής της Επιτροπής του τελευταίους μήνες η ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου τον Ιούνιο του 2018 μαζί και με την αμφίσιμη εκλογική μεταρρύθμιση που δεν σέβεται τις συστάσεις του ODR και της Επιτροπής της Βενετίας είναι διοχτυπητά ε, παραδείγματα της διάβρωσης που λαμβάνει η χώρα τελευταία ε, στην χώρα. Ο σκοπός είναι να εκφοβιστούν τα μέλη της αντιπολίτευσης ε, μαζί και με τη δικαστική εξουσία που παρεμβαίνει στην πολιτική διαδικασία τελικά υποσκάπτεται το κράτος δικαίου. Επιπρόσθετα ε, επιδεινώνεται η ελευθεροτυπία και υπάρχουν επιθέσεις κατά της κοινωνίας των πολιτών. Πέραν όλων αυτών, οι δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου, η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης ε, και η συμμετοχή της κοινωνίας ε, των ε, πολιτών αποτελούν κυρίες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συμπεριληφθεί και στη Συμφωνία με την Μολδαβία. Η κατάχαρση αυτών δεν θα γίνει ανεκτή από αυτό το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό επαναλαμβάνω εδώ αυτό που έχει εκφράσει ήδη το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την πολιτική κρίση του Ιουνίου του 2018 οποιαδήποτε απόφαση για περαιτέρω πληρωμές θα πρέπει να γίνει μόνο όταν έχουν υλοποιηθεί εκλογές βάσει των διεθνών προτύπων στη χώρα. Η Μολδαβική κυβέρνηση μας έχει διαβεβαιώσει για τις θετικές της προθέσεις να βελτιώσει την κατάσταση. Ωστόσο, ε, μία ε, επιτυχής, προκειμένου να έχουμε έναν επιτυχή διάλογο και για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών πρέπει η κυβέρνηση της Μολδαβίας να αναλάβει δράση. Και ήρθε ο καιρό να κρίνουμε την κυβέρνηση της Μολδαβίας βάσει των πραξιών της και όχι βάσει θεωρίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλεκεστάιν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και από τη δική μας την πλευρά να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για το έργο του. Σε πολλά σημεία συμφωνούμε πλήρως όσον αφορά τον δήμαρχο του Κισινάου. Είναι προφανές ότι τα πράγματα δεν ε, είναι σωστά. Έγινε αναφορά και στα βήματα που έχουν σημειωθεί και γι' αυτό θεωρώ ότι δεν θα δυσκολευτούμε να πετύχουμε συμβαστικές ε, λύσεις. Υπάρχουν όμως τρία πράγματα που μας ανησυχούν. Το πρώτο είναι ότι η Επιτροπή της ε, Βενετίας δεν είναι ο Πάπας και εγώ δεν είμαι καθολικός. Και η Επιτροπή της Βενετίας είναι σωστό ότι λέει ποια πρότυπα πρέπει να τηρηθούν, ποιες διαδικασίες θα τηρηθούν, που πρέπει να υπάρξει συνένεση. Αλλά το να πει σε μια χώρα τι εκλογικό σύστημα θα επιλέξει, αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω. Το δεύτερο σημείο είναι γνωρίζετε ότι στην Ολομέλεια δεν κάναμε λόγο για αναστολή της χρηματοδότησης. Αν το κάνουμε όμως, θα πρέπει να το κάνει, να το κάνουμε σωστά και όχι να αφήσουμε μία πίσω πόρτα ανοιχτή που να επιτρέπει ε, κάποιο είδους χρηματοδότηση μέχρι τις εκλογές. Όσον αφορά την ημερομηνία τον εκλογό ώστε να υπάρξει ένα σωστό αποτέλεσμα δεν θα μπορέσουμε μετά να συνεργαστούμε όμως αυτό το μπικοτάζ ε, στις ε, πληρωμές πρέπει να το ε, μελετήσουμε να δούμε πώς θα γίνει. Δεν θέλουμε έμεσα να χρηματοδοτήσουμε τις εκλογές. Το τελευταίο σημείο είναι πιο γενικό και δεν ξέρω αν μπορούμε να το επιλύσουμε σε αυτή την έκθεση. Η... Το αίτημά μας σε αυτούς που 55 απέναντι μας και η εκπλήρωσή του είναι πάντα ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε διαδικασίες διεύρυνσης. Έχουμε δηλαδή την προσδοκία, αλλά δεν λέμε πότε εκπληρώνεται ή όχι. Δεν υπάρχει μια λύση για όλους εδώ, αλλά θα είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητήσουμε με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ κύριε Φλέγγενσταν. Χέλμουτ Σόλτς στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ από την πλευρά μου να, να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή. Συμφωνώ σε πολλά σημεία και τον Ιούνιο. Στην τελευταία συνάντηση είχαμε πολλές σύμφωνες γνώμες, όμως υπάρχουν περίπλοκες ε, διαδικασίες όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Η τελευταία όμως παρατήρηση του κύριου Σανστάιν πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς. και να παρουσιάσουμε γι' αυτό το λόγο τροπολογίες για το θέμα της ε, για την αποκάλυψη, την ενημέρωση του κόσμου για το τραπεζικό σκάνδαλο. Να είμαστε ξεκάθαροι. και να ενημερώσουμε την κοινωνία της Μολδαβίας και να την προωθήσουμε να συμμετάσχει πιο, με πιο δημοκρατικό τρόπο στην ε, μεταρρύθμιση αυτή. Να υπάρξει η παραδοσιακός διαχωρισμός εξουσιών μεταξύ κράτους ε, δικαστικής εξουσίας κτλ ώστε αυτή η λογιστική δομή να σταματήσει να υφίσταται. Έχουμε και το quality report. που είναι σχετικό και με την Ουκρανία, γιατί όταν αυξάνεται η ποιότητα, τότε πάντα αναζωπηρώνεται το θέμα της διαφθοράς και εδώ προκύπτει και πάλι το ερώτημα πώς πρέπει να σταθεί απέναντι σε αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό τη μορφή των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα πρέπει να το εμπολιτήσουμε αυτό το να το ε, μελετήσουμε καλύτερα αυτό το θέμα και να προτείνουμε κατάλληλες ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ. Τελευταία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μία πρόταση μόνο. Άκουσα κάποιους συναδέλφους και μπορώ να πω ότι με τέτοιους φίλους να τους κάνεις τους εχθρούς. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά η Επιτροπή μας απέστειλε αντιπροσωπεία στις αρχές Απριλίου σε Μολδαβία και Ουκρανία και είχα εντολή να ηγηθώ της αντιπροσωπείας και φυσικά και επικεντρωθήκαμε στην υλοποίηση των δύο συμφωνιών και στις δύο χώρες. Ορισμένα σχόλια λοιπόν για το σχέδιο έκθεσή μας. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αστροβίτσιους για την εξαιρετική έκθεση για την υλοποίηση της ε, συμφωνία σύνδεση με τη Μολδαβία. Η υλοποίηση της συμφωνίας και της ε, σε βάθους και σφαιρικής ε, συμφωνίας ελευθερών έχουν απτά αποτελέσματα που έχουν αναφερθεί ήδη. Βελτίωση του χρηματοοικονομικού και τραπεζικού κλάδου και αύξηση του διμερούς εμπορίου. Αναγνωρίζουμε τα βήματα που έχει κάνει η Μολδαβία, όμως είναι σημαντικό να συνεχίσουν οι μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν το 2016 πιο συγκεκριμένα και οι πολιτικές περιποθέσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν που συνδέονται με την θέσπιση αποτελεσματικών δημοκρατικών μηχανισμών. Ένα πολυμερές κοινοβουλευτικό σύστημα, κράτος δικαίου και σεβασμός θεπινών δικαιωμάτων. Είναι σημαντικές προϋποθέσεις για την χορήγηση μικροοικονομικής στήριξης. Με λύπη διαπιστώνουμε ότι μέχρι τώρα η Μολδαβία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές και αυτό οδήγησε στην αναστολή της ε, στήριξη των 100 εκατομμύριων ευρώ. Επίσης, λυπηρό είναι ότι η εκλογική μεταρρύθμιση δεν αντιστοιχεί ε, συστάσεις των δύο επιτροπών, της Επιτροπής της Βενετίας κλπ. Και θεωρώ ότι οποιαδήποτε νέα εξέλιξη θα πρέπει να λάβει χώρα μετά τις προβλεπόμενες βουλευτικές εκλογές και με την προπόθεση ότι θα διεξαχθούν με βάση τα διεθνή πρότυπα. Ναι, ολοκληρώνω, Πρόεδρε. Τέλος. Για το δικαστικό κλάδο, ο τομέας της δικαιοσύνης δυστυχώς ε, δεν ε, έχει περάσει πολλές μεταρρυθμίσεις και εξαιτίας της έλλειψης προόδου θα έπρεπε, μάλλον αναγκάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει τη στήριξή της μέχρι να υπάρξει σημαντική πρόοδος στον τομέα της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έρχεται η σειρά των προσκεκλημένων της Κομισιόν ε, μέσα σε πέντε λεπτά. Θα δώσω το λόγο στον επικεφαλής ε, του τμήματος για την αντιτολική εταιρική σχέση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Um, well, from my side... Και από πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αστροβίτσιους για το εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης που μας έχει παρουσιάσει. Ε, που παρουσιάζει τα πιο βασικά στοιχεία και ε, για την υλοποίηση της Συμφωνίας Σύνθεσης και για τις διμερείς σχέσεις μας με την Μολδαβία. Μετά την ακύρωση των ε, τοπικών εκλογών στο Κισινάου. Τώρα πρέπει να εξετάσουμε ε, τις, ε, τα στοιχεία προβληματισμού που παραμένουν σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου σε σχέση και με την υλοποίηση τη συμφωνία σύνδεση. Ε, και εγώ πιστεύω, συμφωνώ με τον κύριο Φλάκη, αν πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο ακριβεί, αλλά στην περίπτωση Μολδαβία μπορούμε να είμαστε. Και μπορούμε να το συζητήσουμε και δημερό αυτό. Να επισημάνω επίσης ότι η ανησυχία που ε, εκφράζεται στο, στην έκθεσή σας ε, μας βρίσκει και εμάς σύμφωνους και εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια εμείς τα λέμε αυτά ε, στη Μολδαβία, δεν είναι κάτι καινούριο λοιπόν. Τέλος για την εκλογική μεταρρύθμιση. Η θέση που εξέφρασε το Συμβούλιο πρόσφατα παραμένει ίδια και εμείς βλέπουμε ότι δυστυχώς ε, οι συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας δεν ε, λήφθησαν υπόψη. Θα Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε εκ του σύνεγγυς την εκλογική μεταρρύθμιση εδώ σε αυτή την Επιτροπή όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να υπάρχει ε, σωστή παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων του εκλογικού συστήματο κατά τη διάρκεια τη προεκλογική εξαρτία, κατά τη διεξαγωγή των εκλογών και το πιο σημαντικό, μετά τι εκλογέ σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο στη δημοκρατία εν γέννη και στο πολυκομματικό ε, σύστημα πιο ειδικά. Υπάρχει πρόοδο στι ε, οικονομικέ και χρηματοοικονομικέ μεταρρυθμίσει. Βλέπουμε όμω ότι υπάρχει έλλειψη ανεξαρτησίας ε, στη δικαιοσύνη. Αυτό μπορεί να υποσκάψει τις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς και προώθησης του κράτους δικαίου, αλλά μπορεί να υποσκάψει και την οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα της χώρας. Χρειαζόμαστε λοιπόν αμερόληπτη, ανεξάρτητη και υπεύθυνη δικαιοσύνη που να καταπολεμήσει τη διαφθορά, ιδίω ε, στα υψηλά επίπεδα. Αναφέρθηκα στον Ιλαν ε προηγουμένω και ο σεβασμός στο κράτο δικαίου είναι βασικά στοιχεία για την αποκατάσταση της ε, εμπιστοσύνης της κοινή γνώμης της Μολδαβίας ε, στο κράτο και στι δημόσιε αρχές. Έχουμε και μια νέα στρατηγική για τη μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη βάσει και των εμπειριών του παρελθόντος, αλλά το πιο σημαντικό είναι να υλοποιηθούν τα όσα έχουν υιοθετηθεί. Αναφέρθηκε και η έλλειψη προόδου ε, στις έρευνες για τις ε, διαφθορές στον τραπεζικό κλάδο και όπως ανέφεραν και οι Υπουργοί Εξωτερικών Υποθέσεων ε, στο Συμβούλιο το Φεβρουάριο είπαν ότι όλοι οι υπεύθυνοι θα πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη ανεξαρτήτως ε, πολιτικών ε, χρωματισμών και η δημοσιοποίηση της στρατηγικής ανάκτησης ε, δημοσίων περιουσιακών στοιχείων δεν φτάνει γιατί δεν γίνεται όλη η διαδικασία με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Στις 26 Ιουλίου υιοθετήθηκε το πακέτο χρηματοοικονομικής μεταρρύθμισης θεωρούμε ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα κίνδυνο ενομοποίησης παράνομων εσόδων και οι πρώτε πρώτες αντιδράσεις από τους διεθνεί εταίρους δεν είναι θετικές. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις διαδηλώσει που διοργανώνει η αντιπολίτευση που γίνονται με ειρηνικό τρόπο και θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό και να γίνει σεβαστό και από τις ε, μολδαβικές αρχές πρέπει να προστατεύεται το δικαίωμα ε, των ε, πολιτών ε, να διαδηλώνουν ειρηνικά και στον τομέα των μέσων ενημέρωσης. Υπάρχει διάθεση μεταφοράς της σχετικής οδηγίας στο Μολδαβικό Δίκαιο, όμως στην πράξη βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολες συνθήκες για τα μικρά μέσα. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να αποστείλουμε ένα σταθερό μήνυμα προς τις αρχές της Μολδαβίας για να αντιστρέψουμε τις επικίνδυνες τάσεις που παρατηρούνται ε, για την κοινωνία και τη χώρα εν γέννη. Η αιρεσιμότητα, επενθυμίζω, γιατί πολλά μέλη το ανέφεραν, η αιρεσιμότητα για την ε, οικονομική στήριξη παραμένει ένα από τα βασικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να επηρεάσουμε τις ε, αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στη Μολδαβία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στο Λάουρενς Μέρεντιτ που είναι διευθυντής στην ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη ο συνάδελφος αναφέρθηκε στα κύρια σημεία, αλλά συμφωνώ πλήρως με τις παρατηρήσεις τους και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, κύριο Οστροβίτσιος αλλά και την Επιτροπή σας για την εξαιρετική συνεργασία μέχρι την εκπόνηση της ε, έκθεσης αυτή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και πάντοτε θέλουμε να συνεργαζόμαστε, να συνεργαζόμαστε στενά με το Κοινοβούλιο. Το πρώτο σχολείο μου έχει να κάνει με το πόσο σημαντικά είναι αυτά που λέγονται στην πρώτη παράγραφο της έκθεσης, δηλαδή πόσο σημαντική είναι η Συμφωνία Σύνδεσης για τους πολίτες της Μολδαβίας. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου και ότι παράγει αποτελέσματα. Αυτή ήταν μια σημαντική επιλογή που έγινε από το κοινό της Μολδαβίας πριν λίγα χρόνια και νομίζω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πόσο σημαντική είναι η δυναμική αυτής της ε, συμφωνίας ε, να προσφέρει ωφέλη στου πολίτες. Και έχει γίνει πρόοδο ε, προ την επίτευξη των στόχων. των αυτών, φυσικά. Και εμείς συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που εκφράζονται από τον κύριο Στρεβιτσίου και του υπόλοιπου ομιλητέ. Θα ήθελα να επενθυμίσω καταρχήν τη δήλωση της ΥΠΑ της εκπροσώπους και του Επιτρόπου Χάν για την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάο. Υπάρχει μια γραμμή που αντικατοπτρίζει το βαθμό της ανησυχίας. Λέγεται ότι μια, ένα εξάρτητο δικαστικό σώμα ε, ανεξάρτητο από κάθε ποιησή καθώς και ε, δίκες και ανεξάρτητες εκλογές ε, διασφαλίζουν τη δημοκρατία. Έτσι λοιπόν αυτές οι ανησυχίε μα. καταρχήν το δικαστικό σύστημα πρέπει να είναι ανεξάρτητο και δυστυχώς μία από τις πιο δημοφιλείς αποφάσεις που λήθησαν πέρσι είναι ότι, δεν θα πληρώσει ούτε ένα λεπτό από τα 28 εκατομμύρια για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, γιατί θεωρήσαμε ότι τίποτα δεν είχε γίνει για να αιτιολογεί τι πληρωμέ. Δεύτερον, οι εκλογέ, Θέλω να τονίσω δύο τινά. Καταρχήν, ε, οι σοβαρές ανησυχίες ε, που ήδη ανέφερα, ε, τον είπε τον εκπροσώπων της Κοσμισιόν για τις δημοτικές εκλογές του Κεσινάου, αλλά επίσης έχουμε και τις μελλοντικές βουλευτικές εκλογές που θα είναι σημαντική δοκιμή της δημοκρατικής διαδικασίας στη Μολδαβία. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι στο σημερινό περιβάλλον δεν έχει υπάρξει καταρχήν ένα δημοσιονομική υποστήριξη. Ε, όλα ε, ότι όσα υπάρχουν ε, στα έγγραφα ήταν πριν από την τραπεζική κρίση. Επίσης, όλα όσα χρήματα δόθηκαν υποστήριξαν τους πολίτες. Σε ό,τι αφορά τώρα την προεφιστάμενη δημοσιονομική στήριξη, εμείς ε, στο σημερινό περιβάλλον δεν βλέπουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε τις πληρωμέ δεδομένης ε, τη κατάσταση. Ήδη αναφερθήκαμε στη μακροοικονομική βοήθεια. Λοιπόν, θέλω να αναφέρω και δύο άλλα σημαντικά θέματα. Και εγώ συμμερίζομαι τις ανησυχίε που εκφράστηκαν ε, από τα μέλη του Κοινοβουλίου για τις ε, ε, δημοσιονομικέ φορολογικέ μεταρρυθμίσει αλλά και για τη φορολογική αμνηστία. Σε ό,τι αφορά τώρα την τραπεζική απάτη, θέλω να κάνω μια σημαντική διάκριση μεταξύ δύο μερών. Χαίρομαι καταρχήν που λέω ότι υπάρχει, έχει γίνει μία σειρά συστημικών μεταρρυθμίσεων στην δημόσια διοίκηση που πρόκειται να προσφέρουν να ότι ένα τέτοιο περιστατικό δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λαχθέντος αυτούς, όπως είπε και η κυρία Σιμπούλ, πρέπει να απευθυνθούμε στις αρχές προκειμένου να πάρουν περαιτέρω βήματα ε, για την ποινική δίωξη και για την ανάκτηση των πόρων είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Αφενός θεωρούμε ότι έχουν γίνει οι συστημικές μεταρρυθμίσεις, αλλά αφετέρου έχουμε ανησυχίε ω προς τις έρευνες. Ευχαριστώ να απαντήσω σε ερωτήσεις αν τυχόν έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μέρεντι. Να δώσω τώρα τον τελικό λόγο στον εισηγητή. Για να κλείσει το σημείο αυτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εκτιμώ όλα τα σχόλια που ακούστηκαν από τους συναδέλφους και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο συμφωνούν με το σκεπτικό μου κατά την εκπόνηση της έκθεσης. Όντως, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, πολύ ακριβείς. Όταν αυξάνουμε τις προσδοκίες από την πλευρά της Μολδαβίας για την χορήγηση της οικονομικής βοήθειας και από την άλλη τα κριτήρια υπάρχουν ήδη επί χάρτου, αλλά είναι ξεκάθαρα λοιπόν. Αρκεί να ανοίξει κανεί τη σωστή σελίδα και μπορεί να δει τι πρέπει να γίνει και πότε. Και φυσικά εξαρτάται από το επίπεδο τη επίτευξη. από την ποιότητα της επίτευξης. Νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση μας δίνει μια εύρωστη βάση για να βελτιώσουμε την έκθεση και είναι υπομονώ για να έχουμε το τελικό σχέδιο της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Στρεβίτσης. Να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι την επόμενη εβδομάδα στις 7 Σεπτεμβρίου, ώρα 11 το πρωί. Και τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο που είναι η πρώτη εξέταση της έκθεσης που έχει προετοιμάσει ο κ. Μαμίκινς και αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Γεωργία, αλλά η κυρία Μούντι θα μιλήσει εξ του. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Παρουσιάζω λοιπόν την έκθεση εξ ονόματος του συναδέλφου Μάμικινς. Που λέτε τα εξή, αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζω όλοι να περάσετε ωραία το καλοκαίρι. Εγώ προσωπικά αφιέρωσα κατά μέρο τι διακοπέ μου στην ε, συμφωνία με την ε, Γεωργία. Είναι κάτι το οποίο δεν ξεχνώ ούτε κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Ξέρω ότι μόλις χθε ε, λάβατε τις μεταφράσεις, ε, ελπίζω όμως ε, πολλοί από εσάς τουλάχιστον να τη διαβάσατε την έκθεση στα αγγλικά. Είναι η πρώτη έκθεση εφαρμογής για τη Γεωργία και χαίρομαι που καταρτίζεται εκ με τις εκθέσεις για την Ουκρανία και τη Μολδαβία που θα μας βοηθήσει να τις συγκρίνουμε και να έχουμε και προτάσεις βελτίωσης. Οι συμφωνίε σύνδεσης είναι από τα πλέον περίπλοκα ε, διεθνή μέσα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πολύ βασικό για μας είναι ότι βασίζονται σε δεσμευτικές ε, συμφωνίες για την υιοθέτηση ευρωπαϊκών ε, ρυθμιστικών ε, πράξεων. Και αυτό θα ήθελα να τονίσω εδώ. Ο βαθμός της νομικής προσέγγισης θα πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο ε, της αξιολόγησής μας από κοινού και με ποσοτικούς συντελεστές και δείκτες μάλλον. Το 2017 ο στόχος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μπήκε και στο ε, σύνταγμα ε, της Γεωργίας. Ανεξάρτητα λοιπόν από οποιαδήποτε πολιτική αντιπαράθεση. Επιπλέον, προετοίμασαν οι Γεωργιανοί ένα νέο οδικό χάρτη προ την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ελέγξουν όλη την Γεωργιανή νομοθεσία και να εντοπίσουν ε, προσκόμματα προ την προσέγγιση. Ε, και αυτό ήδη υπερβαίνει τις ε, δεσμεύσεις τους ως προς ε, την Συμφωνία Σύνδεσης. Η συμφωνία αυτή είχε πολύ μεγάλες θεσμικές προεκτάσεις για τη Γεωργία και επιβεβαιώνω ότι υπάρχει καλός βαθμός συντονισμού μεταξύ κυβέρνησης και κοινοβουλίου στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο συντονισμός εξακολουθεί να βελτιώνεται ο νομοθετικός προγραμματισμός του Κοινοβουλίου συνάδει πλήρως ε, με το πρόγραμμα της Συμφωνίας Σύνδεσης και η Κοινωνία των Πολιτών ασχολείται και εμπλέκεται ε, στις διαβουλεύσεις. Υπάρχουν θετικές παρενέργειες ε, της Συμφωνίας Σύνδεσης. Αύξηση της οικοδόμησης, εμπιστοσύνη στην κοινή γνώμη και μεγαλύτερη πολιτική ευαισθητοποίηση. Βέβαια υπάρχουν και προκλήσεις. Έλλειψη διοικητικής ικανότητα, ε, δυσκολία προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, ε, καθυστερήσει στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων και έλλειψη πόρων σε ό,τι αφορά την υλοποίηση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εμπλουτιστεί η έκθεση υλοποίηση με περισσότερα κεφάλαια για να αντικατοπτρίζει και τον σφαιρικό χαρακτήρα τη συμφωνία σύνδεση. Ε, προσέθεσα ένα κεφάλαιο για το θεσμικό πλαίσιο και ε, για τον διάλογο μεταξύ λαών και για την ε, συμμετοχή και εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών η Γεωργία εξακολουθεί να ηγείται ε, της ε, ανατολική Τυρκή σχέση και ξέρω ότι υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στη Γεωργία για αυτή την πρώτη έκθεση, γιατί θα δείξει ε, την πρόοδο που έχουν σημειώσει σε σχέση με το ευρωπαϊκό τους όραμα. Και θα ήθελα να συμβάλλετε σε αυτή την προσπάθεια με τις δικές σας απόψει και σχόλια. Τέλος, να κάνω μία πρόταση. Θα ήθελα να πω ότι για να υπάρχει πραγματική προσταθέμενη αξία. Η έκθεσή μας θα πρέπει να στραφεί περισσότερο στην αποτελεσματικότητα της νομικής προσέγγισης με συγκεκριμένους στόχους και να μην ασχολούμαστε μόνο με την εγχώρια πολιτική σκηνή της γεωργίας. Πράγματι, ε, χρειάζεται γεωργία ε, ε ισχυρή ηγεσία για την ε, προσέγγιση της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα, έχουν, τα έχει πάει πολύ καλά η Γεωργία. Υπάρχουν στοιχεία που δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε περαιτέρω σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μούντι και ευχαριστούμε και τον κύριο Μαμίκινς. Ο κύριος Τετίνα, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω τσεχικά Βάλτε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαμίκινς εξουσιοδότηση για τη δουλειά που έκανε για την έκθεση αυτή. Θα ε, ήθελα να πω ότι άκουσα πολύ προσεκτικά τη μελέτη που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο σημείο και αφορούσε την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης με τη Γεωργία. Μπορώ να πω ότι οι επικρίσεις που ακούστηκαν για την πολυφωνία των ΜΜΕ για την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος ε, είναι ε, πάντοτε σημεία που ανακύπτουν και η έκθεση συνάδει με τις δικές μου απόψεις. Έτσι λοιπόν ε, θα ήθελα να ζητήσω να αντικατοπτρίζετε καλύτερη πραγματικότητα στις εκθέσεις αυτές, να εξετάζετε το θέμα του κράτους δικαίου και της διακυβέρνησης και επίσης ε, τι συμβαίνει με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θερμιλιωδών ελευθεριών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ εν μέρη στις πληροφορίες που ακούσαμε, είπα το προηγούμενο σημείο για την έκθεση αυτή, θα ήθελα να πω ότι θα ήταν καλή ιδέα να καλέσουμε τους εκπροσώπους της Εκκλησίας και των θρησκευτικών οργανώσεων εδώ, στη συναντήση μα και από τη Γεωργία και για την Ουκρανία για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε τι δικέ του προσδοκίε. Είναι μέρο τη κοινωνία των πολιτών, άλλωστε. Και έχω και ένα παρόμοιο σχόλιο για τον εξωτερικό διάλογο στη Γεωργία. Εγώ θα καταθέσω και μια σχετική τροπολογία. Θα ήθελα λοιπόν να μου επιτρέψετε να καταθέσω μια διαδικαστική πρόταση από αυτού. Ευχαριστούμε κύριε Γιούρακ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο σε εκπροσώπους της Κομισιόν, ο κύριος Σίβελ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, εκ νέου πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ρόλο του και την αντιπροσωπεία για τη συνεργασία με τη Γεωργία. Αν υπομονούμε για τη συνεδρίαση της ε, επόμενη κοινοβουλευτική επιτροπή που θα λάβει η χώρα στη Γεωργία σε δύο εβδομάδε. Επίση, ε, χαιρετίζουμε την υποστήριξη του γεωργιανού πληθυσμού για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη υποστήριξη που είχαμε σε χώρα της Ανατολικής εταιρική σχέση. Πολλέ φορέ φτάνουμε και στο 80% του πληθυσμού να είναι υπέρ τη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φυσικά διευκολύνει την καλή συνεργασία για την εφαρμογή φιλόδοξη ε, ημερησία διάταξη. Φυσικά η Γεωργία είναι ο πιο φιλόδοξο εταίρο ε, γιατί έχει ουσιαστικά υλοποιήσει τα καθήκοντά της ε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θέλουμε να τονίσουμε ότι επιθυμούμε να ενδυναμώσουμε την πολιτική σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωση με τη Γεωργία. Η Συμφωνία Σύνδεσης έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να ενεργοποιήσει τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ μας. Ε, το τελευταίο Συμβούλιο Σύνδεσης έλαβε χώρα το Φεβρουάριο του 2018 και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γεωργίας ε, τόνισε το πόσο σημαντικό είναι να επιταθεί η περαιτέρω οικονομική ολοκλήρωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αναφέρθηκε η κατάρτιση ενός ε, χάρτη πορείας και φυσικά είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Η υπηρεσία εξωτερική δράση, συνεργασία με την αντιπροσωπεία και με του συναδέλφου τη Κομισιόν, θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη συνεχή εφαρμογή ε, τη σφαιρική και σβάθο ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, ε, καθώ ε, και των ορόσημων για την ε, απελευθέρωση υποχρέωση θεώρηση. Βέβαια, υπάρχουν κάποιε ελλείψει σε κάποιου τομεί συνεργασία. Η απελευθέρωση υποχρέωση θεωρήσεων, η πρώτη αξιολόγηση ήταν θετική. Υπάρχουν όμω κάποιες σημαντικές προκλήσεις που έχουν ανακύψει και εν μέρει έχουν αντιμετωπιστεί. Η γεωργιανή κυβέρνηση έκανε αξιοσημείωτη προσπάθεια να καταπολεμήσει τις ε, καταχρήσεις ε, ε, ό,τι αφορά την απελευθερωμένο ταξίδι από θεωρήσεις έχουμε σημειώσει και πρόεδρο στην εφαρμογή τη φιλική και σβάθο ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργαστεί περαιτέρω με τη Γεωργία ε, σε τομεί όπου χρειάζεται περαιτέρω προσέγγιση, παραδείγματο χάρη δημόσιε συμβάσει, κάποιε τομεί υπηρεσιών, ε, ταχυδρομικέ υπηρεσίε, εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη, ε, ένα σύστημα επιθεώρηση εργασία που να λειτουργεί πλήρω. Εξακολουθούν να υπάρχουν λοιπόν ελλείψει σε αυτού του τομεί. Θέλω να θυμίσω και την ενεργή συμμετοχή της Γεωργίας στην Ανατολική Εταιρική Σχέση είναι και πάρα πολύ ενεργή στη συνεργασία ε, της ΕΠΑ. Έχουν εντοπίσει την ανάγκη να δημιουργήσουν ικανότητες ε, για την προστασία των συνόρων, την αστυνομία και την πολιτική προστασία. Δεν χρειάζεται επίση να το πω, αλλά να επιβεβαιώσω την ε, πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εδαφική κεραιότητα της Γεωργίας και επίσης για τα νομοθετήματα ε, που ε, στοχεύουν σε ένα καλύτερο μέλλον και ε, προσφέρουν στους κατοίκους κάποιες ευκαιρίες ό,τι την κινητικότητα, το εμπόριο και την παιδεία. Από την είπατε εκπρόσωπο υπήρξαν κάποιες δηλώσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει της επαιτίου, της 10 επαιτίου του πολέμου μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας. Ε, θέλουμε να έχουμε ελευθεροτυπία, διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ελεύθερες, ε, ε, ελεύθερο διάλογο για τα θέματα που λειτουργούν και άλλα θέματα που δεν λειτουργούν τόσο καλά όπως είναι τα θέματα του δικοστικού σώματος λοιπά Επίσης αναμένουμε και τις προεδρικές εκλογές που θα λάβουν χώρα το φθινόπωρο να υλοποιηθούν βάσει των διεθνών ε, προτύπων και να μην υπάρξει αντίκτυπος ε, στις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις. Ήδη ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κάπως τεταμένο κλίμα, αλλά ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα μείνουν υπό έλεγχο. Ανεπομονούμε να έχουμε καλή μελλοντική συνεργασία με το μελλοντικό πρόεδρο. Θέλουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μα. Συνολικά όμω συμπεραίνουμε ότι αρκετά καλά τα έχει πάει μέχρι τώρα η Γεωργία και θέλουμε να του υποστηρίξουμε περαιτέρω. Και έχω και την ικανοποίηση να συνοδεύσω τον Επίτροπο Χάν σε λίγε ημέρε στην επίσκεψή του στην Γεωργία. Έχουμε εκεί κάποιε ειδικέ εκδηλώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Um... Αρχικά, να ευχαριστήσω την Κλέρ και την Επιτροπή για την εξαιρετική συνεργασία και την προετοιμασία της έκθεσης. Έχω να πω κάτι παρόμοιο Πρωτίστως βλέπουμε ότι παρέχει ωφέλη στους πολίτες η Συμφωνία Σύνδεσης και γι' αυτό είναι σημαντικό να μην τα θεωρούμε δεδομένα. Η πολιτική κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Πριν από μερικά χρόνια ήταν μια μεγάλη επιλογή κατεύθυνση για την ε, Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία και είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι υπάρχουν απτά ωφέλη για τους πολίτες Συμφωνούμε ότι η Γεωργία τα πάει καλύτερα από τις υπόλοιπες χώρες. Βλέπουμε αύξηση του εμπορίου, οικονομικές ευκαιρίες για επενδυτές έξω από την Ουκρανία, θεσμικές αλλαγές, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και η Συμφωνία Σύνδεσης και η εφαρμογή θα προσφέρει ωφέλη στο σύνολο των πολιτών. Και αυτό μπορώ να το συνδέσω και με την αναφορά στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας, γιατί είναι πολύ σημαντικό α, σημείο αυτό. Σχηματίζει την κοινή γνώμη η Εκκλησία. Πολύ από τους, ένας από τους παραγωγούς μελιού από τη Γεωργία, και χάρη στη συμφωνία σύνδεση μπορούν πλέον να το πουλήσουν στο Lidl τη γειτονιά μου. Είναι λοιπόν σημαντικό σημείο γιατί όταν ο κόσμος βλέπει ότι μπορεί πραγματικά ε, να ωφεληθεί στην καθημερινή του ζωή τότε θεωρώ ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε το του διάλογο. Ε, το θεωρώ σημαντικό. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε το πρώτο σχολείο Ανατολικής Γειτονίας. Πολύ σημαντική εξέλιξη που δείχνει την ε, διάθεσή μας να επενδύσουμε στον ανθρώπινο δυναμικό, να επενδύσουμε στην νεολαία. Ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και σε αυτό. Να μην έχουμε όμως την εντύπωση ότι όλοι είναι ρόδινα Υπάρχουν κάποιες βασικές προκλήσεις που πρέπει να σημειώσουμε. Η δικαιοσύνη και πάλι. Υπήρξε αναστάτωση στις αρχές του καλοκαιριού το να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη οι πολίτε σε ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα είναι βασικό και πρέπει να λάβουμε μέτρα γι' αυτό. Όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές, θα πρέπει οι εκλογές να γίνονται με έναν ελεύθερο δημοκρατικό τρόπο. Θα τις παρακολουθήσουμε στενά, γιατί είναι ένα, μια σημαντική στιγμή. Επίσης το φθινόπωρο θα έχουμε μια σημαντική συνάντηση με την κυβέρνηση. 25 Νοεμβρίου συνάντηση με το Κολέγιο των Επιτρόπων μετά την επίσκεψη του πρόεδρου Γιούνκερ το καλοκαίρι. Εδώ δείχνει τη δέσμευση, φαίνεται η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην γεωργία και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να ε, προχωρήσουν και να προωθήσουν ε, την εφαρμογή της συμφωνίας με έναν εντυπωσιακό θα έλεγα τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε θα ξαναδώσουμε το λόγο στην κυρία Μούντι. Ευχαριστώ. στην Επιτροπή και στην Επίση Εξωτερική Δράση. Τα σχόλια σα για τη συνεχιζόμενη εμπλοκή σα θα πω πρώτα ότι δεν εξαρτάται από εμά να έχουμε εσωτερικού πολέμου με τον πληθυσμό της Γεωργία. και αυτό με επαναφέρει σε βασικά στοιχεία που ε, ε, αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι. Η σημασία του έργου μας στη Συμφωνία Σύνδεσης είναι ο αντίκτυπος που θα έχει στο λαό και στα ωφέλη που θα επιφέρει στο λαό. Αυτό θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της δουλειάς μας και γι' αυτό μπλεκόμαστε τόσο εντατικά σε αυτό το πρόγραμμα. Ένα... Ε, αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στη διαδικασία επικοινωνίας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, για τη συμμετοχή τους και σε εσά Ανυπομονώ να συνεργαστούμε και στο μέλλον και για την επόμενη συνεδρίση PSA ε, το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μούντι. Να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεση των προλογιών είναι επίσης στις 7 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί. Τώρα, το τελευταίο σημείο είναι το σχέδιο έκθεσης που έχει ετοιμάσει ο κύριος Γκάλερ σχετικά με την εφαρμογή Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας και να δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλερ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, πριν από μερικές μέρες η Ουκρανία είχε την εθνική της γιορτή χρειάστηκε χρόνια για να αναπτύξει και να συντηρήσει την εθνική της ταυτότητα Ουκρανία. Αυτή είναι η συνέπεια των προηγούμενων επιρροών που είχε και είναι κατανοητό ότι χρειάζεται μια διαδικασία διαφο... Ε, καθάρισης ως προς το μοντέλο εξέλιξης που θα ακολουθήσει η Ουκρανία και ποιο θα είναι το επίκεντρο, πώς θα κινηθεί μάλλον η χώρα σε σχέση με την Ευρώπη. Μετά την δημοκρατική επαναστασία ε, πριν από 14 χρόνια ε, υπήρξαν εξελίξεις, αλλά δυστυχώς έπρεπε ε, να υπερασπίστον αυτή της Ουκρανία ενάντια σε, στην στρατιωτική επίθεση της γειτονικής Ρωσίας. Συνεχίζει να υπάρχει ανησυχία σε αυτό το θέμα. Δέχεται επιθέσεις από τους γείτονες στη μέση της Ευρώπης μπροστά στα μάτια μας. Βρίσκεται σε στενή σύνδεση πλέον ε, με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμφωνία και η απελευθέρωση των θεωρήσεων είναι ξεκάθαρα σημάδια. Συναντήσεις συχνές λαμβάνουν χώρα με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας πριν από τέσσερα χρόνια ε, αποφασίσαμε και για μια σφαιρική σε βάθο ζώνη ελευθέρων συναλλαγών και με, αφού τεθεί πλήρω ε, σε εφαρμογή αυτή η συμφωνία προτείνω ότι ε, μπορούμε να κλείσουμε ένα θετικό συμπέρασμα γιατί έχει καταφέρει να σημειώσει πρόοδος προς την ευρωπαϊκή ένταξη. Υπάρχουν όμως ακόμα κάποιες βασικές ανησυχίες και προκλήσεις κυρίως όσον αφορά την δικαιοσύνη, την αποκέντρωση, την ενέργεια, την υγεία, τη συντάξει, την εκπαίδευση. Υπάρχουν ε, βέβαια και κάποιες θετικές εξελίξεις. Ε, η είδηση δικαστηρίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την οικονομική διαφάνεια. Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για την αποκέντρωση Υπάρχουν λυπή μέτρα για την ε, αποδυνάμωση του ολιγαρχικού κράτους. Χρειάζεται να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα και πλέον θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και στα εξή σημεία. Ε, η δήλωση που πόθεν έσχεσαι από ε, μέλη, ε, μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων η δημιουργία, η ταχεία δημιουργία και στελέχωση του ανώτου δικαστηρίου για την καταπολέμηση διαφορά. Αυτά είναι βασικά για την εφαρμογή της συμφωνίας και από την πλευρά της Ουκρανίας και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δημιουργηθεί αντιστοίχως και η οικοδόμηση ικανοτήτων στο διοικητικό κομμάτι να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία και να την υποστηρίξουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ουκρανία συμπληρώνει ένα χρόνο από, την, ε, προ... Ε, από, την, από ε, τις τελευταίες εκλογές. Παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ανησυχία τη στάση των πολιτών, την υποστήριξη που είχαν πριν από τέσσερα χρόνια ως ε, ε, ψηφοφόροι για την εξυγχρονισμό της χώρας. Βλέπουμε ότι όλα αυτά πλέον αντικαθίστανται από την απογοήτευση που έχουν για τις άθλιες οικονομικές συνθήκες διαβίωσης και για τις, ε, την έλλειψη αλλαγών στην κρατική διαφθορά. δεν μπορούν επίσης να κατανοήσουν τις πρόοδους που γίνονται, γιατί δεν επεξηγούνται με σωστό τρόπο. Είναι σημαντικό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίε για τους πολίτες, να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και να υποστηρίξουμε τον κύκλο της μεταρρύθμισης. Το στενό πλαίσιο της εκθέσης δεν μας έδωσε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε όλα τα σημεία και σε όλες τις εξέλιξεις των τελευταίων χρόνων. Θα είναι επομένως και άλλα στοιχεία, αλλά κυρίως θα ήθελα να αναφερθώ ε, στην ε, ε, κλοπή που γίνεται εις βάρος των φυσικών πόρων το πώς παρεμποδίζονται οι κοινοτικές εκλογές κάτι που θεωρώ δικαιολόγητο καθώς και το θέμα που υπάρχει στον τομέα τη αποκέντρωση. Αναμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλερ. Ο κύριο Γιούρακ έχει το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Μου αρέσουν τα βασικά στοιχεία και η δομή της έκθεσης. περιέχονται λεπτομεριστικά για την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας, όμως έχω να κάνω ένα σχόλιο για το άρθρο 20 αυτή της ε, έκθεσης. Θα πρέπει η Ουκρανία να επικυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Αυτό είναι σύμφωνο με τους στόχους της Επιτροπής, αλλά δεν είναι συμβατό με τη συνθήκη συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι, που δηλώνουν ότι δεν θα ε, εμπλακεί ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κατηγορίες θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν είναι αυταπόδεικτο να επιμένουμε σε πράγματα τα οποία είναι αντιφατικά στα δικά μας κρατημέλη. Παραδείγματο χάρη, όσον αφορά το στεγματικό δικαστήριο της Βουλγαρίας στην προηγούμενη Προεδρία, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε σε αντιπαράθεση με το βουλγαρικό σύνταγμα. Δεν θα πρέπει να προωθούμε σε εξωτερικό επίπεδο να επιμένουμε σε ιδεολογικές αλλαγές. Θα πρέπει να σεβαγόμαστε την ελευθερία των εθνών, γιατί η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να έχει τη δική της άποψη για το τι είναι καλό για το Lodge, το ίδιο που, θα έκανε, που έκανε και η Βουλγαρία. Άρα να προσέχουμε ότι μιλάμε ε, για ένα θέμα που ακόμα είναι συζήτηση στα δικά μας κράτη-μέλη και γι' αυτό θα πρέπει να επιβάλλουμε πράγματα στην ε, Ουκρανία. Όσον αφορά την προστασία των κοινωνικών μειονοτήτων, γνωρίζουμε ότι η Ουκρανία είχε μια βασανισμένη ιστορία υπό την Σοβιετική κατοχή. Πολλοί που ζούσαν ε, στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης εκτοπίστηκαν αλλού και αντιστρόφως. Αυτό δημιούργησε πολλές δυσκολίες. Σκέφτομαι π.χ. την, ε, την ε, ρωμακαθολική μειονότητα στο Ελβίβ. Αυτή η κοινότητα έχει ήδη λάβει μέτρα για να προστατέψει τον εαυτό της, όμως υπάρχουν ακόμα προβλήματα με τα δικαιώματα και την προστασία τους, γιατί δεν συμφωνούν, παραδείγματο χάρη, με αποφάσεις ε, του Δήμου το 2010, όπου αποφάσισαν μία από τις πιο πολύτιμες ε, ε, εκκλησίες στην ε, Ευρώπη να χρησιμοποιηθεί ως συνευλιακός χώρος. Θα πρέπει η εκκλησία να καθορίσει το πώς θα χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν τέτοιου είδους θέματα, να καταδικάζουμε τέτοιες αποφάσεις, γιατί η αλλαγή μπορεί να ενισχύσει τον πλουραλισμό και την αμοιβαία, τον αμοιβαίο κοινωνικό σεβασμό. Γι' αυτό θα ήθελα να το λάβετε και αυτό υπόψη στην έκθεσή σας και να το ενσωματώσετε με έναν κατάλληλο τρόπο. Ευχαριστούμε. Κύριε Γιούρεκο, ο κύριος Βαλές έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστήσω τον κύριο Γκάλερ που μας ε, παρουσίασε μια ισορροπημένη ε, έκθεση και πολύ ακριβή. Εγώ ως εισηγητής ε, της ΙΝΤΑ θέλω να υπογραμμίσω ότι η γνωμοδότηση περιλαμβάνει όχι μόνο τις εμπορικές πτυχές αλλά και πολιτικές πτυχές που θα μπορούσαν να ε, να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την, το ανοιχτό και δίκαιο εμπόριο με όλου του εταίρου. Η Ουκρανία είναι ένας από τους πιο στενούς εταίρου μα ε, στο εμπόριο και θέλουμε να λειτουργήσει η συνεργασία σφαιρική και βάθος ε, Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών ε, ισχύει από την 1η-1η 2016 και είναι τμήμα ευρύτερης συμφωνίας σύνδεσης ε, τη οποία οι διατάξει έχουν εφαρμοστεί προσωρινά από τον Νοέμβριο του 2014 από τη Σκοπιά τη Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Τονίζω την ανάγκη και τα δύο μέρη να ανοίξουν αμοιβαία τι αγορέ του για αγαθά και υπηρεσίε που βασίζονται σε προβλεπόμενου κανόνε η συμφωνία θέλει να προωθήσει το εμπόριο σε αγαθά και υπηρεσίες μεταξύ της Ένωσης και της Ουκρανίας μειώνοντα σταδιακά του δεσμού ε, και ευθυγραμμίζοντα του κανόνε τη Ουκρανία ε, με του κανόνε Ευρωπαϊκή Ένωση σε αγιορικά προϊόντα και βιομηχανικού τομεί. Έτσι λοιπόν, καλωσορίζουμε την αύξηση στου εμπορικού όγκου μεταξύ Ένωση και Ουκρανία σε βαθμό που η διαφοροποίηση των εξαγών τη Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τονίζεται η κανονιστική προσέγγιση μεταξύ Ένωσης και Ουκρανίας είναι να ένα στο εργαλείο που φέρνει την Ουκρανία πιο κοντά στην Οικονομική Ένωση και συνεισφέρει στη διευκόλυνση του εμπορίου σε καλύτερο επιχειρηματικό κλίμα και σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ουκρανίας. Επίσης, δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι η DCFTA είναι μέρος της διαδικασίας μεταρρύθμισης βάσει της καλής διακυβέρνησης και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία της συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας για την επιβολή κυρώσεων ε, σε σχέση με την Κρυμαία και την Ανατολική Ουκρανία. Τέτοιες κυρώσεις ε, θα αυξήσουν την πίεση προκειμένου να έχουμε μια ειρηνική επίλυση των εδαφικών προκλήσεων της Ουκρανίας. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η Βερχόφνα Ράντα πρώτη ανάγνωση οθέτησε το νομοσχέδιο για την προστασία των Ουκρανικών ε, δασών καθώς είχαμε ένα μεγάλο εμπορικό φραγμό στον τομέα αυτό. Θέλω επίσης να αναφερθώ σε ένα θέμα που ανησυχεί πολύ και ήταν ε, θέμα ε, εκτεταμένης δημοσιογραφικής έρευνας ε, τα ορυχεία στην περιοχή των Μπάς. Περιμένω γραπτή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα, όμως εν το μεταξύ θέλω να δηλώσω ότι λόγω κυρώσεων ε, έχουν ε, παγώσει ε, τα περιουσιακά στοιχεία ορισμένων. Υπάρχει ουσιαστικά ρύθμιση από την κυβέρνηση των αποκαλούμενων δημοκρατιών. Η φυσική πόροι είναι αντικείμενο εκμετάλλευση εταιριών που έχουν εθνικοποιηθεί και ελέγχονται από διαφορετικέ κυβερνήσει. Η ρώτησή μου λοιπόν στην Κομισιόν είναι αν η αγορά και η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτών των φυσικών πόρων ε, που ε, προέρχονται από τις επαρτιστικές δημοκρατίες θα πρέπει να επιτρέπεται. Γνωρίζουμε ότι ο κάθε κέρδος από αυτές τις πωλήσει ή εξαγωγές έμεσα ή άμεσα ε, ωφελούν τις αποσχιστικές δημοκρατίες και τις κυβερνήσεις τους. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή τη διάσταση. Ευχαριστούμε κύριε Βαλέσα. Ο κύριος Σέλμπερ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα και εγώ θα ήθελα ε, να σε τον κύριο Γκάλερ για την εξαιρετική αυτή η έκθεση. Πληρέστατο το κείμενο, παρότι πράγματι μπορούν να προσθεθούν κάποια νομοθετικά στοιχεία. Είναι όμως πολύ καλό το σχέδιο έκθεσης και θα ήθελα να σταθώ και στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Επιτροπής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, και του κυρίου Γκάλερ και με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων εν γέννη. Είναι πολύ χρήσιμη και γόνιμη αυτή η συνεργασία και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι. Και νομίζω ότι και για τη Συμφωνία σύνδεση. η Σχετική Επιτροπή κάνει πολύ καλή δουλειά για την ε, υλοποίηση της Συμφωνίας. Πολύ θετική είναι και η οικοδόμηση δυναμικού που γίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό τον Pat Cox για την ε, βελτίωση της ε, νομοθετικής ικανότητας, που είναι και γνώστης εξάλλου της ουκρανικής πραγματικότητας. Η αντιπροσωπεία μας στο Κίεβο εργάζεται άοκνα για τη μεταφορά του ενωσιακού κεκτημένου στην ε, Ουκρανική νομοθεσία στις Βρυξέλλες. Η υλοποίηση της εφαρμογής είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε πολύ στενά και εμείς και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και θεωρούμε ότι επί της έχει αυξήσει τις προσπάθειές της ε, η κυβέρνηση με την υιοθέτηση ενός ε, σχεδίου δράσης για τη Συμφωνία Σύνδεσης και με την υιοθέτηση μια σειράς μηχανισμών ε, και με μια σειρά διευκολύνσεις στις διαδικασίες νομοθετικών πράξεων. Κατά τη διάρκεια τη επίσκεψη τη ΕΠΑ τη εκπροσώπου στην Ουκρανία τον Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ξεκίνησε και μια εκστρατεία ενημέρωση. Προχωρούμε μπροστά μαζί ε, που μιλάει για τα απτά αποτελέσματα της Συμφωνίας Σύνδεσης και μιλάει και για το θεματολόγιο αλλαγών και μεταρρυθμίσεων δεν άκουσα πολλά για αυτή την ε, καμπάνια. Είναι κάτι όμως το οποίο θα πρέπει να έχουμε κατά νου και για την Ουκρανία αλλά και για τη Μολδαβία και τη Γεωργία. Για να εξηγούμε καλύτερα ε, ποιο είναι το όφελος ε, των συμφωνιών αυτών για τους πολίτες. Επομένω, αναγνωρίζουμε τις, την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα, αλλά όπω είπε και ο εισηγητή, πολλά ακόμα μένουν να γίνουν. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και τα μελλοντικά φιλόδοξα βήματα θα πρέπει πάντα να εντάσσονται ε, στο, στη Συμφωνία Σύνδεσης. Τομείς προτεραιότητας, καταπολέμηση διαφθοράς, ε, φυσικά και βρίσκεται στην κορυφή ε, των προτεραιοτήτων. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι θεσπίστηκε ανακοινώθηκε η θέσπιση ενός ε, δικαστηρίου για την καταβλέμηση της διαφθοράς ε, που θα συνδέεται και με το Εθνικό Γραφείο, την Εθνική Υπηρεσία Καταβολέμησης Διαφθοράς και με τον ε, Ισαγγελέα Διαφθοράς. Είναι σημαντικό να μην υπόκειται σε καμία επιρροή αυτό το δικαστήριο και ο εισαγγελέα πρέπει να ενισχυθεί και να λάβει την απαραίτητη στήριξη αυτό ο θεσμό. Υπήρχαν κάποια προβλήματα το καλοκαίρι, μπορεί να τα έχετε παρακολουθήσει κι εσείς. Βέβαια υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωση τη Ουκρανία. τα ανέφερε και ο κύριος Γκάλαρ και άλλοι συνάδελφοι, βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και διαφάνεια σε πολλού τομεί. Εν ώψη των ε, εκλογών το Μάρτιο και το φθινόπωρο του 19 υπάρχει ένα σαφές μήνυμα ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια μεταρρυθμίσεων. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να σταματήσουν τώρα οι προσπάθειες μεταρρυθμίσεων και να μπουν όλοι ε, σε κλίμα προεκλογικό. Δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Τέλος, για την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία της κυριαρχίας, εμείς είμαστε ξεκάθαροι και αμετάκλητοι στη στήριξή μας ως προς αυτό. Το μερικό άνοιγμα της γέφυρας Κάσπιν από δύο, δύο μήνες και οι αυξανόμενες εντάσεις στη θάλασσα Αζόφ είναι ανησυχητικές εξελίξεις. Και ο Λέξεν Σόφ τώρα βλέπουμε ότι εδώ και πάνω από 100 μέρες κάνει απεργία πείνας. Εμείς έχουμε απευθύνει πολυάριθμες εκκλήσεις για την απελευθέρωσή του και ελπίζουμε οι ρωσικές αρχές να μας ακούσουν ε, και να κάνουν αυτή την ε, δήλωση, την κίνηση καλής θέλησης. Και πρόσφατα και η ε, καγκελάριος Μέρκελ συνομίλησε με τον Ρώσο πρόεδρο. Θα μας επιτρέψει ενδεχομένω αυτό να προχωρήσουμε λίγο, γιατί σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωση και από πλευρά Ουκρανία περιμένουμε τον νόμο για το ηθικό καθεστώ των ε, κατεχόμενων περιοχών που θα πρέπει να επεκταθεί τον Οκτώβριο και είναι μία από τι προποθέσει ε, από εδώ και πέρα και για την υλοποίηση τη συμφωνία του Μίνσκ. Τέλος, ε, εμπόριο από τις ε, αποσχισμένες περιοχές. Εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα του εμπορίου, αλλά όπου υπάρχει σφραγίδα των Ουκρανικών τελωνίων, έχουμε την εντύπωση ότι πρόκειται για Ουκρανικό προϊόν. Αν έχετε λοιπόν ε, συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιων προϊόντων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε και τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπάρνερ που είναι επικεφαλής ε, της ομάδας υποστήριξης στην Ουκρανία. Ευχαριστώ. Προσθέσω να μιλήσω γερμανικά. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ και τους υπόλοιπους για τις εκθέσεις που έδειξαν ότι, ότι στην εκτίμηση της κατάστασης και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ουκρανία συμφωνούμε ως επιτοπλίστων και ευχαριστούμε και για τις εκθέσεις και για τις ε, συζητήσεις που γίνονται και για το γεγονός ότι είναι πολύ περιεκτικές και έχουν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωκοινοβουλίου επίσης. Υπάρχει επίσης μεγάλη κατανόηση και αυτό φαίνεται στην έκθεση ποια είναι τα διαφορετικά επίπεδα επίπεδα προβλημάτων ε, στην Ουκρανία που πρέπει να μας απασχολήσουν. Ε, έγινε λόγος για τις ε, προκλήσεις μεγάλες, την επιθετικότητα της Ρωσίας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι τα πάντα το θέμα αυτό με τη Ρωσία. Θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλουμε ώστε και μακροοικονομικά να σταθεροποιηθεί το κάναμε τα περασμένα έτη, θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Κατά δεύτερον, η ομάδα στήριξης ε, για την Ουκρανία και ο ρόλος της ε, θα κάνουμε λόγο για institution και capacity building, οικοδόμηση ικανοτήτων. Μιλήσαμε και για άλλε χώρε σχετικά με αυτό το θέμα. Έχουμε λοιπόν τη δημόσια διοίκηση, η οποία πολλέ φορέ είναι υπερβολικά φορτισμένη, όχι μόνο να εκπονήσει νομοθεσίε, αλλά και να του εφαρμόσει. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία τρία χρόνια ε, 3 εκατομμύρια ευρώ σε μέτρα στήριξης και σε μια έκθεση από κοινού και με άλλους εταίρους κάνει λόγο για την αποκέντρωση που είναι σημαντικό στοιχείο. Αυτό που εν μέρη αναφέρθηκε στην έκθεση είναι ότι πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση της διοίκησης και παράλληλα φάνηκε στην έκθεση ότι είμαστε πρωτοστάτες ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, στήριξη για την κοινωνία των πολιτών, για την καταπολέμηση της θωράς. Και φυσικά υπάρχει και ο τρίτος τομέας για την Συμφωνία Σύνδεσης. Από κοινού στους διάφορους τομείς, αλλά και με τα Υπουργεία μελετήσαμε την πρόοδο προς την εφαρμογή της ε, συμφωνίας. Σημαντικό είναι πώς θα συνεχίσουμε στον τομέα αυτό με την παρακολούθηση και την εκπόνηση εκθέσεων συμφέρουμε με τις συστάσεις και όσον αφορά το capacity building είναι σύμφωνα και με τις συστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε πριν τις εκλογές για να συνεχιστούν οι προσπάθειες μεταρρυθμίσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά από την πλευρά μας. Ε, προς στιγμή δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε κύριε Βάκνερ. Ο κύριος Γκάλερ για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την στήριξη της γενικής γραμμής που ακολουθούμε και για όλους που συμμετέχουν, που εμπλέκονται από την Επίσης εξωτερική δράση και από την Επιτροπή και από την πλευρά μου. Υποστηρίζω αυτά που είπατε για τους πολιτικούς κρατούμενους στη Ρωσία. Θα πρέπει να το φέρουμε το θέμα στο φως της δημοσιότητας. Στο διάλογο που γίνεται στο πλαίσιο αυτών των εκθέσεων. ένα συνάδελφος τόλμησε να πει ότι κάνουμε λόγο για τρία αποτυχημένα κράτη, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και αυτός είναι ο συνάδελφος που συνεχίζει να κάνει τις δηλώσεις ε, γιατί θεωρεί ότι δεν έχουν προχωρήσει αρκετά αυτές τις τρεις χώρες στην δημοκράτηση και γενικά δεν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Η Ρωσία βέβαια χρειάζεται αυτές τι ολιγαρχίες εκεί. Δεν ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε ολιγάρχες στο Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο και με το καταστημένο Είμαστε υπέρ στην πλευρά των μεταρρυθμίσεων που θα εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες. Και να οργανωθεί η κοινωνία με έναν επιτυχή τρόπο. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε σε αυτό το ύφο. Ευχαριστούμε κυρία Γκάλερ. Ευχαριστούμε και τους υπόλοιπους ομιλητές. 3 ε, Σεπτεμβρίου, ε, συγγνώμη, 7 Σεπτεμβρίου είναι πάλι η κατάθεση τροπολογιών. Ο κύριος Οστρεβίτσιος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω μια μικρή δήλωση για πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Καμπότζη. Όπως ε, γνωρίζετε, Κιμ Σόχα από την αντιπολιτευσή παραμένει στη φυλακή και το Εθνικό Κόμμα Διάσωσης Καμπότση είναι εκτός ε, νόμου. Επιβλήθηκαν ε, κυρώσεις στην ελευθερία γενικές εκλογές του Ιουλίου χωρίς πραγματικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης να μπορούν να έχουν ε, συμμετάσχει. Ε, πήρε το κυβερνών κόμμα 125 θέσεις από τις 125 έδρας. από τις 125 απευθύνουμε έκκληση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την Κομισιόν συγκεκριμένα, να παρουσιάσει στην Επιτροπή μας την έκθεση της ε, διερευνητικής αποστολής που έλαβε χώρα στα μέσα του έτους. Πρωτοφανής πολιτική κρίση, καταστολή της αντιπολίτευσης ε, πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να απαντήσουμε μια κατάλληλη γραμμή πολιτικής. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη σχέση μας με την Καμπότζη ως συνήθως, καθώς η δημοκρατία στην Καμπότζη είναι σε κίνδυνο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Οστρεβίτσιους. Έχουμε καταγράψει τη θέση σας. Ολοκληρώνουμε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Η επόμενη συνεδρίαση θα είναι στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 από τις 3 το μεσημέρι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς ε, και χαίρομαι που ολοκληρώθηκε ο αγώνας τους. Ε, ελπίζω να έχουν γίνει δεκτές οι προτάσεις τους για τις συνθήκες εργασίας. Σας ευχαριστώ.